I have told you I have my opinion. I think it's for to say. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die... Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρία τη Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού και έχετε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Ρωτώ εάν έχετε ενστάσει καταρχάς. Όχι, άρα εγκρίνεται. Η συνεδρία εξάγεται δημοσία. Υπάρχει η διερμηνία στις συνήθεις γλώσσες. Και μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου η συνεδρία. Και έτσι περνώ στο σημείο 3 της της διάταξης, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 9η Ιανουαρίου, 20-21 Ιανουαρίου, 22 Ιανουαρίου, 23 Ιανουαρίου και ρωτώ εάν υπάρχουν προτάσεις για τροποποίηση των πρακτικών. Όχι. Εγκρίνονται. Σημείο 4 στην της διάταξη. Εδώ έχουμε την ακρόαση του υποψηφίου μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η συγγήτρια είναι η κυρία Αιάλα Σέντερ και επί τη ευκαιρία καλωσορίζω τον προτινόμενο υποψήφιο για το ελεγκτικό συνέδριο από την Αυστριακή Κυβέρνηση, κύριο Όσκαρ Χέριξ. Καλώς ήρθατε. Ε, βεβαίως, ο μεγαλύτερη είναι τόσο λιγότερο και οι βουλευτές που έρχονται. Ίσως θα μπορούσα να γεμίσω και ένα βιβλίο από τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις μου από την υπηρεσία μου ως Προέδρου με το θέμα αυτό. Αλλά ίσως το γεγονός ότι είναι μεγάλη αίθουσα και είναι πιο απλωμένοι οι βουλευτές μπορεί να καλυφθεί με, την, με τα οργανωτικά μας. Η συγκήτρια λοιπόν να μας κάνει μια μικρή παρατήρηση, μια μικρή εισήγηση με τις παρατηρήσεις της. Έχουμε μια σειρά από γραπτές ερωτήσεις αποστήλη, τις έχετε απαντήσει. Κύριε Χέριξ, παρακαλώ λάβετε το λόγο για να συνεχίσουμε με τη συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή ε, Ελέγχου του Προπολογισμού, θα ήθελα να ξεκινήσω στα αγγλικά την παρουσίασή μου και εν συνεχεία να απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα στι ερωτήσει σα. Στα γερμανικά δηλαδή, για να μπορώ να είμαι πιο ακριβή στι απαντήσει μου. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας συστηθώ και να ε, έρθω αυτοπροσώπως στην Επιτροπή σας, ε, την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, μετά τον ορισμό μου για να συμμετάσχω ως μέλος στο ελεγκτικό συνέδριο. Το πρώτο θέμα της παρουσίασής μου είναι η εμπειρία μου στον τομέα του λογιστικού ελέγχου. Έχω εργαστεί για περισσότερο από 22 χρόνια στο Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο και ενεργά διενήργησα πάνω από 100 ελέγχους επιδόσεων σε τομείς ε, ομοσπονδιακής διοίκησης αλλά και διοίκηση επίπεδο κρατήριο ε, ενέργεια, μεταφορές, ε, περιβάλλον, γεωργία, έρευνα, οικονομικές επιδοτήσεις, απασχόληση και επίσης διενέργησε ελέγχου σε κρατικές επιχειρήσεις όπως η Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας ή ο Εθνικός Ρωτηλοπτικός Φορέας της χώρας μου. Στο πλαίσιο λοιπόν των ελέγχων αυτών θα ήθελα να σας δώσω έμφαση σε ελέγχους που άπτονται άμεσα του τομέα των δημοσίων οικονομικών, των επενδύσεων της διαχείρισης κινδύνου. Κατ' εμέ η πεμπτουσία για, μια για έναν αποτελεσματικό έλεγχο δεν είναι μόνο η τήρηση ε, των ε, κριτηρίων και οι μετρήσεις που προκύπτουν από τους ελέγχους για να είναι δυνατόν ε, τα κεφάλαια των φορολογμένων να αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένας από τους βασικούς στόχους μου λοιπόν θα είναι αυτός ως ε, επίδοξο μέλος του Ευρωπαϊκού Ελληνικτικού Συνεδρίου. Το δεύτερο σημείο. Ε, χρηματοοικονομική διαχείριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουν και επικεφαλής ε, ε, των ζητημάτων που αφορούσαν τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασχολήθηκα λοιπόν με τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάφερα με τις προσπάθειές μου να έχω μια σημαντική συμβούλη ε, στην διασφάλιση ποιότητας της χρηματοοικονομικής διαχείρισης ε, στην Αυστρία και ιδίως στον τομέα της κοινή διαχείρισης στηρίζοντας ταυτόχρονα τις δραστηριότητες και την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στους ελέγχους που διενήργησε στην ε, Αυστρία. Εν των νέων μέτρων για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιομικής πολιτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο συντονισμός και η συνεργασία ε, των ανώτατων ελεκτικών φορέων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δημιουργεί μια νέα πολύ σημαντική διάσταση προς την πρόκληση αυτή. Έχω λοιπόν την αντίληψη ότι η συντονισμένη αυτή συνεργασία θα καταστήσει το δικό μου έργο ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελληνικτικού Συνεδρίου και πολύ σημαντικό. Επίσης, κατά την άποψή μου, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει αποφασιστικά να στρέψει την προσοχή του στη διενέργεια περισσότερων ελέγχων επιδόσεων, ελέγχων απόδοσης. Αυτή η πεποίθηση μου βασίζεται στην εμπειρία μου στον τομέα των λογιστικών ελέγχων. Διότι τα αποτελέσματα των ελέγχων είδα ότι οδήγησαν σε αποδοτική, αποτελεσματική χρήση των δημοσίων κονδυλίων. Κατόπιν τούτου, οι χαράκτες πολιτικής όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα πρέπει αφενός στο μέλλον να είναι σε θέση να έχουν στη θέση τους δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου να διατυπώνουν αποτελεσματικές στάσεις, ξεκάθαρη στάση για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Και επανέρχομαι, ε, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία και στη συνεργασία με τα ομοσπονδιακά και κρατηδιακά κοινοβούλια που θα με βοηθήσει. Τρίτο σημείο, ανεξαρτησία οι υπάλληλοι του ελεκτικού συνεδρίου θα πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα και να μην υπάρχει ουδεμία αμφιβολία για την ε, ανεξαρτησία τους, ε, την αμεροληψία τους, την ακαιρεότητά τους και να δίνουν συνεχώς πρέπει ε, αποδείξεις τούτων των ιδιωτήτων για να δείχνουν ότι είναι η δράση τους επαγγελματική και οι έλεγχοι που κάνουν είναι επαγγελματικοί και αμερόληπτοι με βάση τα διεθνώς, διεθνώς ε, αποδεκτές αρχές σε κάθε ένα από τα λειτουργήματα που ίσκησα έδρασα σύμφωνα με τις πεπιθήσεις μου και όταν ασκούσα τα καθήκοντά μου ως ε, ελεγκτής βασίστηκα πάντοτε ε, και πρόσεξε ιδιαίτερα τα πολύ λεπτά θέματα Είμαι λοιπόν ουσιαστικά ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, ε, έχω σημαντική ε, επαγγελματική εμπειρία και βέβαια ακαδημαϊκές γνώσεις ε, και πήρα στη δημόσια λογιστική, στις δημόσιους ελέγχους. Η μέχρι τώρα σταδιοδρομία μου εστιάστηκε απολύτως στον τομέα του ελέγχου και τη βελτίωση των δημόσιων συστημάτων. Θα επιθυμούσα λοιπόν να συνεχίσω ε, την ίδια δράση σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο για να διευκολύνω και να ενισχύσω τη στενή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινόβουλου και ιδιαίτερα με την Επιτροπή σας, Στην Επιτροπή Ελέγχου του Με Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος Τόερερ, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Θα παρακαλέσω τώρα την η συγγήτρια να λάβει το λόγο και θα ακολουθήσουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω τον κύριο Χέριξ, τον Αυστριακό υποψήφιο. Υποψήφιο μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου. Φυσικά και έχετε ένα εξαιρετικό βιογραφικό, έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και σημαντικά προσόντα ακριβώ στους τομείς με τους οποίους ασχολείται το ελεγκτικό συνέδριο. Έχετε ιδίω εμπειρία στους ελέγχους ως ελεγκτής, αλλά με ενδιαφέρουν πολύ και τα προσόντα που διαθέτετε σε ό,τι αφορά την παροχή συμβουλών και ε, τη διεξαγωγή συνεχούς διαλόγου με το Αυστρακό Κοινοβούλιο για τη βελτίωση του ομοσπονδιακού και του τοπικού επίπεδου, συνεργασία με το ομοσπονδιακό και τοπικά κοινοβούλια. Ήθελα να σας θέσω το εξή ερώτημα. Σχολιάσατε μεταξύ άλλων κάτι που θεωρούμε σημαντικό. σε σχέση με το το πρόγραμμα του ελεγκτικού συνεδρίου, την εμπειρία αυτή και το πολιτικό πρόγραμμα ενό κοινοβουλίου, βλέπετε να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Εμείς δεν θα θέλαμε να ε, υπάρξουν παραδείγματα αναποτελεσματικότητας που δυστυχώς τα είδαμε, διότι ορισμένες από τις γνωμοδοτήσεις ή ε, ελεγχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου έφτασαν καθυστερημένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δεν αντικατόπτριζαν το άμεσο πολιτικό ε, ενδιαφέρον και στο Κοινοβούλιο θέλαμε πάρα πολύ μια γνωμοδότηση του ελεκτρικού Συνεδρίου. Χωρί βέβαια να απολέσετε την αυτονομία σα και την ανεξαρτησία σα, πώ βλέπετε ε, το ενδεχόμενο να μπορέσετε να συνεργαστείτε και πάντοτε σε επαφή με την επικαιρότητα και τι ανάγκε ε, τη νομοθετική εξουσία. Ποια θα είναι η σχέση με το Κοινοβούλιο. Επόμενο ερώτημα. Έχετε μακρά εμπειρία στο Αυστριακό Ελεκτικό Συνέδριο. αλλά είπατε ότι είχατε εμπειρία και από το τι γίνεται στο, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό ε, Συνέδριο. Υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή σε σχέση με την αύξηση αυτή της συνεργασίας που κατά ανάγκη ε, είναι μια πραγματικότητα, το είδαμε και με τις τράπεζες αυτό. Και υπάρχει ανάγκη λοιπόν τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεργάζονται πιο στενά. Όλα αυτά όμω ανοίγουν και μια συζήτηση. Υπάρχουν κάποιοι που όπω εμεί συμφωνούν, συμφωνούμε απόλυτα ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να ενισχυθεί ω θεσμικό όργανο και θα πρέπει οι υπόλοιποι να συνεργάζονται στου τομεί βέβαια που είναι απαραίτητο με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Υπάρχει λοιπόν μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει σε σχέση με το κατά πόσον θα έχουμε ένα είδος δικτύου εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων, που όμως ενδεχομένως να αποδυναμώσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας άποψη από αυτού. Από τις απαντήσεις σας που έμαθα και πολλά πρέπει να σας πω, ε, από τις απαντήσεις λοιπόν στο ερωτηματολόγιο, νομίζω ότι η θέση σας είναι πιο πολύ να ενισχυθούν, να ενισχυθεί το ελεγκτικό συνέδριο. Επίσης μιλάτε για το κόστος ε, των ελέγχων, κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όταν μας δώσετε λοιπόν τις απαντήσεις σας, ε, θα είναι μεταξύ των αρμοδιοτήτων και ευθυνών σας ε, ή μάλλον ήταν στο, στις αρμοδιότητες σας στο Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες απαιτήσει για ελέγχους και όλο και μεγαλύτερο είναι το κόστος, διότι είναι πιο πολύπλοκη και πιο ευρύς αυτή η έλεγχη αυξάνεται το κόστος ενώ μειώνονται και οι προπολογισμοί. Πώς θα εξασφαλίσουμε λοιπόν έναν πάρα πολύ καλό έλεγχο μέχρι το τελευταίο σέντ, αλλά και έναν αποτελεσματικό ε, έλεγχο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή σας, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, στο μηχανισμό ελέγχου των τραπεζών, διάσωση των τραπεζών, και τη θέση σας ε, ενδεχομένως στο νέο μηχανισμό. Αυτό το Συμβούλιο Ελεγκτών που προβλέπετε, ποια είναι η άποψή σας, το άτομο που θα εκπροσωπεί το ελεγκτικό συνέδριο, θα έχει ευθύνη, θα λογοδοτεί, από ό,τι φαίνεται ούτε μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε μπροστά στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ποια είναι η δική σας άποψη η παρουσία του ελεγκτικού συνεδρίου στον οργανισμό αυτό δεν θα πρέπει να είναι απλά ατομική παρουσία, αλλά θα πρέπει να έχει και μια θεσμική ιδιότητα το, το όργανο αυτό. Είπατε για κάποια έκθεση που έγινε μέσα σε 10 μήνες, μήνες συγγνώμη παραδειγματική έλεγχη. Πώς επιτυγχάνετε το, την ισορροπία μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεσματικότητας των ελέγχων. Διότι συχνά εδώ βλέπουμε ε, να μην ε, δίνονται οι πόροι που απαιτεί ή ζητά το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να του δίνουμε το παρέτο ανθρώπινο δυναμικό, του ζητάμε περισσότερα και περισσότερους ελέγχους. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε. Εγώ θα προτείνω κύριε υποψήφιε να συγκεντρώσουμε και άλλες ερωτήσεις και επομένως ας ε, δώσω το λόγο τώρα στην ε, συντονίστρια του Λαϊκού Κόμματος κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Μας ικανοποιεί που πρόκειται υποψήφιος από Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο με σημαντική πείρα Παρακαλώ να μας εξηγήσετε πού βλέπετε τις προτεραιότητες στην συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως γνωρίζετε από το εθνικό επίπεδο, λειτουργεί αυτή η συνεργασία μεταξύ βουλών και συνεδρίων και στο εθνικό επίπεδο. Πού μπορούμε να ρίξουμε το βάρος μας εδώ, έτσι ώστε να ενισχύσουμε το ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου. Εμείς έχουμε και κάποιες, κάποια σημεία κριτικής, για παράδειγμα την διάρκεια του, που χρειάζεται το, Ευρω... το ελεγκτικό συνέδριο για την εκπόνηση ειδικών εκθέσεων. Φαίνεται ότι υπάρχουν κανόνες εσωτερικών διαδικασιών του ελεγκτικού συνεδρίου που εμποδίζουν τα μέλη του να συντάξουν ταχύτερα τις σχετικές εκθέσεις. στο Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο τι συζητείτε σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και προσοχή στις απαντήσεις σας γιατί τα γνωρίζουμε ήδη αυτά. Δεν ξέρω, θέλετε να ακούσετε την επίσημη ή την ανεπίσημη εκδοχή, κυρία συνάδελφε, ρωτάω ο πρόεδρος. Εσείς, κύριε Γκάιερ, τώρα τον... Α, δεν παρετείτε. Ο κύριος Μούλντερ. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Ήδη είναι εντυπωσιακή η εμπειρία του υποψηφίου στο Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ολίγες γενικές ερωτήσεις. Ένα σημαντικό γεγονός στην ετήσια ζωή του Κοινοβουλίου είναι η υποβολή της εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εμείς εξετάζουμε κάθε φορά το ποσοστό, ποσοστό σφάλματος στη γενική εκτέλεση του κανονισμού. Τα τελευταία τρία χρόνια υπήρξε κάπως υψηλότερο και αυτό δεν ικανοποιεί το Κοινοβούλιο όμως όλα βασίζονται στην υπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι η δήλωση αξιοπιστίας μπορεί να δοθεί μόνο όταν το ποσοστό σφάλματος δεν υπερβαίνει το 2%. Τα τελευταία 9 χρόνια δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο 2%. Θεωρεί ο υποψήφιος ότι το 2% είναι ρεαλιστικός στόχος, εξακολουθεί να είναι ρεαλιστικός στόχος. 2% στην εκτέλεση του αυστριακού προϋπολογισμού. Είναι ρεαλιστικό. Αν έχετε κατέβει και παρακάτω θα ήθελα να το μάθω. Γι' αυτό ρωτώ. Η υπόθεση του 2% είναι ρεαλιστική. Και βεβαίω, όπω έχετε πει και στι γραπτέ σα απαντήσει, πάντοτε υπάρχει σχέση μεταξύ κόστους και ωφελία. Μήπως το κόστος των ελέγχων θα γίνει υπερβολικά υψηλό εφόσον επιμείνουμε στο 2%. Δεύτερη ερώτηση. Για ένα θέμα ιδιαίτερα δημοφιλές εδώ στο Κοινοβούλιο. Στην κοινή διαχείριση νομίζομαι ότι υπάρχει τελικά έλλειψη ευθύνης από πλευρά των χωρών μελών. Δεν αντιλαμβάνονται οι χώρες μέλη δηλαδή ότι τελικώς είναι υπόλογες. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμένει στο να γίνεται στο αρμόδιο πολιτικό επίπεδο δήλωση αξιοπιστίας που να λέει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού στη συγκεκριμένη χώρα μέλος έγινε σύμφωνα με τους κανόνες. Τώρα υπάρχουν και ορισμένες ενστάσεις και ιδίω από τις χώρες εκείνες μέλη που έχουν ομοσπονδιακή οργάνωση. Γι' αυτό και ρωτώ, στην περίπτωση της Αυστρίας θεωρείτε ότι θα είναι δυνατόν να φτάσουμε σε αυτή την δήλωση αξιοπιστίας του κράτους μέλους, ναι ή όχι. Ευχαριστώ, Γιάννη. Η κυρία Αντρεάσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Έριξ για τις ε, γνώσεις και την εμπειρία του που δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους με την κατάλληλη πείρα ώστε να οριστούν μέλη του Ελεκτικού συνεδρίου προκειμένου να είναι σε θέση να ε, εγκρίνουν τις δαπάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς λέτε ότι δεν ε, στρέφεστε μόνο προς την ορθότητα των δαπανών αλλά σας ενδιαφέρει και το όφελος ή η επιτυχία καλύτερα ενός προγράμματος που διεξάγεται και χρηματοδοτείται από τα χρήματα του Ευρωπαίου Προλογίου. Όπως ξέρετε το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει εκδώσει βεβαίωση για να βεβαιώσει την νομιμότητα των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελευταία 19 χρόνια. Άρα εάν δεν μπορεί να βεβαιώσει την νομιμότητα και το τυπικό, την τήρηση των κανόνων, πώς μπορεί να επαληθεύσει και τη διεξαγωγή των προγραμμάτων. Ευχαριστώ, κύριος Ιρνχάους. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχω αρμοδιότητα στις ε, δύσκολες ερωτήσεις εδώ. Η ανεξαρτησία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Προβλέπετε Υπάρχουν ε, κάποιες αναφορές από τον ε, τύπο της Αυστρίας, ημερήσιο και περιοδικό, τις οποίες ασφαλώς θα έχετε λάβει υπόψη και ίσως θα πρέπει να συνοψίσω τους αδέλφους για να τους εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. Ο κύριος Σπίντλεκε, μέλος, ε, πρόεδρος του FVP, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Αυστρία, έχει εκτεθεί σε επικρίσεις που φτάνουν ακόμη και στα έδρανα του δικού του κόμματος μετά τις εκλογές φαίνεται ότι η πορεία του κόμματος αυτού θα είναι κακή, θα χάσει ως και τη θέση του στο κόμμα. Και φαίνεται, από ό,τι λένε τουλάχιστον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο τύπος να ε, θέλει να, λάβει, να πάρει τη θέση να διαδεχθεί τον κύριο Χάν ως επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ίσως ο κύριος Βέγκεμπάουρ να πάρει τη θέση του, φίλος του κυρίου Σπιντλέκε, όπου φαίνεται πως έχει ήδη ξεκινήσει με την ε, κυρία Σπιντλέκε που έχει λάβει θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτά τουλάχιστον λένε τα κουτσομπολιά στον τύπο. Ίσως είναι όλα αυτά κάπως αφηρημένα, αλλά η ε, πολιτική αυτή που δεξάγεται χάρη σε φιλίες φαίνεται να λειτουργεί ακόμη καλά στην Αυστρία. Και ασφαλώς τέτοιου είδους επικρίσεις και ερωτήσεις θα κληθείτε και εσείς να απαντήσετε. Είστε λοιπόν φίλος και εσείς προσωπικός του κύριου Σπίντλακε, επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος και Υπουργού των Οικονομικών και επίσης έχετε σκοπό να αναλάβετε συνέχεια κάποιες θέσεις ε, ουσιαστικές, ε, αποφασιστικές στην Αυστρία και ενδεχομένω και στην Επιτροπή. Και επίσης, η κυρία Σπίντλακε είναι όντως ε, μέλος του δικού σας επιτελείου αυτή τη στιγμή. Τρίτον, Υπάρχει όντως αλήθεια στους ισχυρισμούς ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακρόαση στο, Εθνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίθετα με τα όσα προβλέπουν οι παραδόσεις και τα έθιμα και επίσης μπορείτε, νομίζω, ότι μπορείτε να εκπληρώσετε το, το ρόλο σας με αυτούς τους όρους. Ο Πρόεδρος, πολλές ερωτήσεις. Ήθελα να δώσω το έργο και στον κύριο Μπέρμαν αλλά ίσως είναι καλύτερο να ακούσουμε πρώτα απαντήσεις. Μετά, μετά εσείς, μετά. Α, καλά, ο κύριος Μπέρμαν λοιπόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Το Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο κάνει ελέγχους απόδοσης επιδόσεων πέραν των δημοσιονομικών ε, σε σχέση με τις πολιτικές που εκτελούνται στην Αυστρία θα γνωρίζετε φαντάζομαι ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναπτύξει ελέγχους όχι μόνο δημοσιονομικούς αλλά και επιδόσεων. Έλεγχο διαχείρισης, ούτως είπε. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο αυτό σε όλους τους τομείς πολιτικής, δηλαδή δεν είναι εύκολο να πτυχθούν αυτή η ελεγχή απόδοση από το ελεγκτικό συνέδριο. Εσείς τι νομίζετε ότι θα χρειαστεί το ελεγκτικό συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να επιτελέσει και αυτό το έργο των ελέγχων ε, διαχείρισης ή ε, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση αποτελεσματικά. Πώς αναλύετε εσείς αυτήν την κατάσταση και το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Πολύ σύντομα κυρία Γκέκλε. Θα ήθελα να πω στον κύριο Έρεν Χάουσερ ότι εγώ έχω άλλη αντίληψη της υπόθεσης αυτής ή είναι ευέλικτος ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι ειδήσει στον αυστριακό τύπο ή τι να σας πω. Εγώ την ιστορία με αυτή την ε, κυρία Σπίντλεκε την έχω ακούσει ως ότι χρειάστηκε να ε, φύγει από τη θέση της. Ότι θα, θα, θα, πρέπει να φύγετε εσείς για να έρθει η κυρία Σπίντλεκε, θα σας αντικαταστήσει δηλαδή. Θα θέλατε λοιπόν να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις παραπάνω. Ευχαριστώ. Δεν φανταζόμουν ότι η σημερινή συνεδρίαση θα έπαιρνε τέτοια συναρπαστική τροπή. Παρακαλώ και περιμένω μεγάλη αγωνία της απαντήσεις. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Δύσκολες ερωτήσεις μου θέσατε και πολλές. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες και θα αρχίσω με την πρώτη της εισηγήτριας. Η, τι δουλειά έχει το ελεγκτικό συνέδριο στα πολιτικά προγράμματα των κοινοβουλίων. Εδώ πρέπει πρωτίστως να εξετάσει κανείς ότι τα ελεγκτικά συνέδρια και το ευρωπαϊκό έχουν κάποια καθήκοντα να εκπληρώσουν. Καθήκοντα που έχουν ρυθμιστεί στις συνθήκες, καθαρά ότι το ελεγκτικό συνέδριο συμβάλλει στον έλεγχο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στηρίζοντας το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Εδώ πρέπει κανείς να κινήσει από την αφετηρία ότι οι ελεγκτές λαμβάνουν τους πολιτικούς στόχους ως μέτρο. Καθήκον μας δεν είναι να ασκήσουμε πολιτική ούτε να λάβουμε πολιτικές αποφάσεις. Καθήκον μας είναι να εξετάσουμε την εκτέλεση των στόχων με βάση τις πολιτικές αποφάσεις. Αυτό νομίζω μπορούμε να το πράξουμε και καλά. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένε προϋποθέσεις. Πρώτον, οι στόχοι πρέπει να είναι καθορισμένοι. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι στόχοι, συχνά εμείς εν ελήψη στόχων βάλαμε benchmark. Κοιτάξαμε δηλαδή στην Αυστρία ποιες είναι ανάλογες επιδόσεις σε άλλους τομείς. Ή κάναμε και συγκρίσεις με την αλλοδαπή. Πού μπορούμε δηλαδή να επιτύχουμε την μέγιστη απόδοση. Δεύτερο, ο παράγων χρόνος. Για τους ελέγχους και για τις εκθέσεις είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη εκτός από την ποιότητα που πρέπει να είναι η απαιτούμενη, να είναι και επίκαιρε εκθέσεις. Τι νόημα έχει, και αυτό βεβαίως άπτεται και του δικού σας έργου, να έρθουν με καθυστέρηση οι εκθέσεις, όταν ήδη έχουν ληφθεί οι πολιτικές αποφάσεις. Παράδειγμα από τη δική μου εμπειρία στην πράξη. Εξετάσαμε, για παράδειγμα, την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών και κάναμε κρίσιμες συστάσεις για την εποπτεία των τραπεζών και ασφαλιών στην Αυστρία. Κάναμε ορισμένες κρίσιμες και κριτικές συστάσεις, επειδή όμως στόχος μας ήταν, διότι τότε ετοιμαζόταν νομοθέτημα στην Αυστριακή Βουλή, Στόχος μας ήταν να είμαστε απολύτως επίκαιροι. Μέσα σε 9,5 μήνες ετοιμάσαμε την έκθεση και την υποβάλαμε στην Εθνική Βουλή και οι συστάσεις που περιλάβαμε ήταν στη βάση μοντέλων και αποτέλεσαν την βάση για το κυβερνητικό νομοσχέδιο. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι το ιδεώδες. Δεν θα είναι πάντοτε δυνατόν να εφαρμοστεί, αλλά ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να προσφέρουμε και ποιότητα αλλά και να είμαστε και έγκαιροι. Μιλήσατε μετά για την συζήτηση με τις τράπεζες και την συνεργασία με τις ελεγκτικές αρχές και το ελεγκτικό συνέδριο και την ενδεχόμενη δημιουργία ενός δικτύου. Και βάλατε μέσα και το στοιχείο του κόστους των ελέγχων. γιατί τη συνεργασία γενικά πρέπει να πω ότι είμαι πεπισμένος ότι οι δημόσιοι έλεγχοι δεν μπορούν να περιορίζονται από τα σύνορα. Χρειάζεται λοιπόν ένα δίκτυο των ελεγκτικών αρχών και υπερεθνικά σε επίπεδο ένωσης, αλλά και στο επίπεδο των κρατών μελών που να περνάει και στις περιφέρειες. Πρέπει να επιτύχουμε, και αυτό είναι έτοιμα για όλους μας και για τα ελεγκτικά συνέδρια, να αρθούμε στο ύψος της αποτελεσματικότητας. Δηλαδή πρέπει με όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Αυτό είχε εύκολα, αλλά είναι δύσκολο να γίνει. Υπάρχουν διάφοροι τομείς όπου μπορούν να επιτεθούν βελτιώσεις. Θα επανέλθω σε αυτά απαντώντας και σε άλλες ερωτήσεις για το θέμα της κοινή διαχείρισης, για παράδειγμα, που είπε ο κ. Μίλτερ. Έχουμε εδώ και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και νομίζω και σε αυτό αναφέρθηκε ο κ. Βουλευτής. Κυρίε και κύριοι, γνωρίζετε ότι εδώ ιδρύθηκε ένας μηχανισμός για να στηρίξει τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Μιλούμε για ποσό Τη τάξη των 700 δισεκατομμυρίων ευρώ και από αυτά 18 δισεκατομμύρια πρέπει να καταπληθούν ήδη και αυτά είναι χρήματα των χωρών μελών τελικά δηλαδή των φορολογουμένων. Στο αρχικό σύμφωνο δεν προβλεπόταν ούτε ο παραμικρός εξωτερικός έλεγχος, παρά μόνο από ελεγκτές της ιδιωτικής οικονομίας, που σίγουρα είναι σημαντικός. Αλλά τελικά σε βάση πρωτοβουλίας του Γερμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου και το Αυστριακό συμμετέσχει αμέσω, και εγώ μάλιστα ήμουν και επικεφαλής αντιπροσωπείας που μετέβη από την Αυστρία στη Γερμανία, και προσπαθήσαμε με πολλές συζητήσεις να υποβάλουμε προτάσεις που όλο και βελτιώναμε μέχρι να επιτύχουμε να δημιουργηθεί ένας οικονομικός έλεγχος σε ένα όργανο πενταμελές από τους ανώτατους ελεγκτές των ε, χωρών μελών και από μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου, του ευρωπαϊκού δηλαδή. Και δεν έχουμε φτάσει στο τέλος εδώ, δεν έχουμε φτάσει τον απόδοτο στόχο, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και σημαντικές ελλείψεις, διότι οι εκθέσεις που συντάσσει το Συμβούλιο υποβάλλονται μόνο στον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ή στο Συμβούλιο Διοικητών των Τραπεζών και όχι στο ελεγκτικό συνέδριο. Δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση αυτή, διότι δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια. Όμως, μη λησμονείτε ότι ξεκινήσαμε από το μηδέν και το αποτέλεσμα είναι ήδη σημαντικό. Πρέπει ωστόσο να μην φυστούμε προσπαθειών για να το βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω. Τώρα για το κόστος των ελέγχων. Και αυτό έχει σχέση με την αποτελεσματικότητα και την ένταση. Αποτελεσματικότητα και ένταση των ελέγχων σημαίνουν κόστος. Δεν έχει όμως νόημα να αυξάνουμε το κόστος διαρκώς για να διορίζουμε και άλλους ελεγκτές. Θα γνωρίζετε την καμπύλη αυτή, την διαδρομή της καμπύλης, όπου στο τελευταίο της τμήμα ανέρχεται πάρα πολύ αργά. Όσο και όσα και μέσα να διαθέτεται, η βελτίωση της αξιοπιστίας είναι πάρα πολύ περιορισμένη στο τέλος της καμπύλης. Άρα το στοιχείο του κόστους πρέπει κανείς να το έχει διαρκώς προοφθαλμών και να υπάρχει μια σχέση μεταξύ κόστους και ωφέλειας. Δεν μπορώ να σας δώσω την συνταγή που θα λύσει όλα τα προβλήματα, πρέπει να το δει κανείς αναπερίπτωση. Τρίτη ερώτηση. Καλύτερος έλεγχος μέχρι το τελευταίο λεπτό του ευρώ. Εγώ νομίζω δεν απαραίτητο αυτό. Σημαντικό είναι η ελεγκτική δραστηριότητα να ελέγχει πρωτίστως τα συστήματα, τις λειτουργίες. Να δούμε πού υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν τα, οι ελεκτρικοί μηχανισμοί, υπάρχει ε, διαφανές σύστημα υποβολή εκθέσεων. Αυτά είναι σημαντικά. Εάν διαπιστώσουμε λοιπόν στη διαδρομή αυτή ότι υπάρχουν ελλείψεις που μας ανησυχούν, τότε είναι σημαντικό να προχωρήσουμε ένα επίπεδο πιο κάτω και να ελέγξουμε πιο συγκεκριμένα ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, τι γίνεται με το ποσοτικό στοιχείο. Όμως, όπως και με το ποσοστό σφάλματος, κανένας έλεγχος δεν μπορεί να φτάσει στο μηδέν, στο ποσοστό μηδέν, διότι πρέπει δίπλα σε κάθε υπάλληλο να κάθεται και ένας ελεγκτής. για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Κυρία Εισηγητρία, εγώ συμπλήρωσα λίγο την ερώτησή σας. Βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα και εγώ συμφωνώ ότι ο εκπρόσωπος του, συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ασφαλώς οφείλει να αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και για την ε, περίπτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, όπως είπα πριν, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, η έκθεση που συντάσσει το ε, Συμβούλιο Διοικητών πηγαίνει στο Συμβούλιο και δεν πηγαίνει στο Κοινοβούλιο. Εγώ θα προσπαθήσω ενδεχομένως και σε διαπραγματεύσεις με τις χώρες μέλη να συμβάλλω στην επίτευξη κάποιων βελτιώσεων. Άλλη ερώτηση, ανθρώπινη πόρη και οικονομική απόδοση. Και στο Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουμε θέσει κάτι επανάληψη το θέμα. Αν εξετάσει κανείς την οργανωτική δομή του Αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα διαπιστώσει ότι κάθε 3-4 χρόνια επανεξετάζουμε τη δομή μας. Είχαμε ένα τμήμα γεωργικών ελέγχων ιδίω οικονομικών γεωργικών ελέγχων. Είδαμε τώρα ότι με την ενίσχυση των χρηματοδοτικών οργάνων της Ένωσης χρειάστηκε να ενισχύσουμε περισσότερο το τμήμα ευρωπαϊκών οικονομικών ελέγχων. Να δώσουμε δηλαδή πολύ μεγαλύτερο βάρος σε αυτά. Και να συμβάλλουμε σε μια ευαισθητοποίηση για την διαχείριση του προϋπολογισμού, του ευρωπαϊκού ενωσιακού προϋπολογισμού δηλαδή, μέχρι και τις περιφέρειες της ε, χώρας μας. Από το Κοινοβουλίο λαμβάνουμε συνεχώς νέες εντολές. Από, από, το, από το Κοινοβούλιο μας λαμβάνουμε νέες εντολές ως ελεγκτικό συνέδριο. Για παράδειγμα, μας ανέθεσαν τώρα να ελέγχουμε και τις τοπικές κοινότητες. Παλαιότερα είχαμε στην αρμοδιότητά μας 24 κοινότητες. Καταφέραμε με εντατική προβολή της επιχειρηματολογίας να μειώσουμε τον αριθμό των κατοίκων των ε, κοινοτήτων που καλούμασταν να ε, ελέγξουμε, να κατέβει δηλαδή, επομένως φτάσαμε από τις 24 κοινότητες στις 70 κοινότητες που ελέγχουμε. Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να βελτιώσουμε την απόδοση των οικονομικών ελέγχων. Έχω σημειώσει και στο βιογραφικό μου. Επί 7 χρόνια είχα και παράλληλη δραστηριότητα ως ελεγκτής και τον εσωτερικό έλεγχο των δομών του ε, Αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ξεκινήσαμε ανάλυση δική μας, στο όργανό μας, για να ελέγξουμε το χρόνο που χρειάζονταν οι εκθέσεις μας για να εκπονηθούν και οι έλεγχοι μας για να διεξαχθούν. Και η γραμμή μας είναι αυτή. Αυτά ως απαντήσεις για την κυρία Αγιάρα Σέντερ. Τώρα, η κυρία Κρέσλε προτεραιότητε μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ελεκτικού Συνεδρίου και τι βελτιώσει μπορεί να επιτύχει κανείς. Το ερώτημα έθεσα και εγώ σε αυτόν. Περισσότερες, περισσότερη έλεγχη αποδόσεων. Εμείς στην Αυστρία κατεξοχήν διεξάγουμε οικονομικούς ελέγχους. Αυτό έχει σχέση και με την ιδιαιτερότητα που έχουμε στη χώρα μας, αν και μπορούμε να το συζητήσουμε ήδη από τώρα αυτό, ότι το Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο κάνει και την συνολική έκθεση για το ομοσπονδιακό επίπεδο. Το financial statement δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών και όλων των Υπουργείων. Εμείς όμως συντάσσουμε την έκθεση. Δηλαδή εμείς σχολιάζουμε και αξιολογούμε και τις αποκλήσεις από τον προϋπολογισμό. Εξετάζουμε τις συνθήκες πλαίσια, πώς έχουν, σε ε, αν έχουν οδηγήσει ενδεχομένως σε καθυστερήσεις και αναλύουμε και συγκεκριμένους τομείς πολιτικής που συνεπάγονται σημαντικό κόστος, για παράδειγμα συντάξεις, κοινωνική στέγη κλπ. Είναι διαφορετική η θέση του Αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου βέβαια από αυτήν του Ευρωπαϊκού. Εμείς διεξάγουμε και τους ελέγχους αξιοπιστίας. Διότι δεν κάνουμε εμείς δήλωση αξιοπιστίας, το statement of assurance, εφόσον διαπιστώσουμε ελλείψεις, τότε υπάρχει μια διαδικασία όπου καλούμε τις αρμόδιες αρχές, τα Υπουργεία δηλαδή, να διορθώσουν τις ελλείψεις που έχουμε εντοπίσει. Μπορούμε να ασκήσουμε λοιπόν σημαντική επιρροή για τις βελτιώσεις αυτές. Τι εννοώ με λίγα λόγια. Κάτι μπορεί να βοηθήσει εσά το έργο σας. Η δήλωση της αξιοπιστίας, εφόσον δεν την έχετε αυτήν, στην έκθεση, την ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο διότι διέπεται και από την ε, συνθήκη της λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί κανείς να σκεφτεί εάν τις διαπιστώσεις αυτές για την νομιμότητα εάν μπορούν να εμπλουτιστούν και με ένα στοιχείο σκοπιμότητας. Δηλαδή, μία δαπάνη η οποία ελέγχεται και εφόσον θεωρηθεί ότι σωστά έγινε και σωστά αποδόθηκαν οι λογαριασμοί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου της νομιμότητας. Όμως ίσως αυτό να μην σας αρκεί, διότι δεν γνωρίζετε για ποιο λόγο έγινε η σχετική δαπάνη. Τι επέτυχε. Δημιουργήθηκαν κάποιες ε, θέσεις απασχόλησης, δημιουργήθηκε κάποια αξία. Πώς ελέγχθηκαν οι δαπάνες και οι επιπτώσεις αυτές. Ίσως αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί το στοιχείο αυτό της σκοπιμότητας δηλαδή. Εγώ δεν μιλώ εδώ για διαζευτικό δίλημα, είτε το ένα είτε το άλλο, να γίνει είτε το ένα είτε το άλλο. Να γίνει περισσότερο μια μετακίνηση προς performance audit. Νομίζω ότι αυτό θα βελτιώσει και την ποιότητα της δικής σας εργασίας. Και κάτι που εγώ θεωρώ σημαντικό και το Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ότι οι ελεγκτές σημειώνουν και κριτικές παρατηρήσεις. Εγώ το έθεσα ως στόχο και αυτός θα ήταν και στόχος μου εδώ. Δεν μπορεί να υπάρχει σημείο κριτικής που να μην συνοδεύεται από σύσταση. Δεν αρκεί οι ελεγκτές να ασκούν κριτική. Θα έρθετε εσείς και θα με ρωτήσετε μετά, ε, ωραία, και μετά τι να κάνουμε, πώς να το καταφέρουμε καλύτερα. Βεβαίω, οι ελεγκτέ δεν μπορούν να τα γνωρίζουν, δεν μπορούν να γνωρίζουν τα πάντα. Οφείλουν όμω να σκεφτούν να υποδείξουν και τρόπους για την καλύτερη διαχείριση των δαπανών. Εδώ μπαίνει και το στοιχείο της ποιότητας. Για, για παράδειγμα, για το πρόγραμμα εργασιών. Πόσα performance audits θα πρέπει να κάνει. 25 το 2012, τώρα πάλι 24, 25 πόσο, μήπως χρειάζεται περισσότερα. Εγώ θα έλεγα όμως ότι αποφασιστική δεν είναι η ποσότητα, όσο η ποιότητα. Το περιεχόμενο των εκθέσεων που θα λάβετε και οι συστάσεις που θα περιέχουν, ώστε να σας βοηθήσουν στο έργο σας. Τώρα για το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα για το τι γράφεται στην Αυστρία για το ελεγκτικό συνέδριο. Δύσκολο να απαντήσω. Εμείς στο ελεγκτικό συνέδριο το αυστριακό δηλαδή συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το ευρωπαϊκό και αυτό έχει σχέση με το ότι για κάθε έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου τον συνοδεύουμε και εμείς εφόσον γίνεται στην Αυστρία πάντοτε είναι παρόν και ένας ελεγκτής δικός μας που παρακολουθεί. Παρακολουθεί με ποιον τρόπο εργάζεται το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνεδρίο. Και ενδεχομένως αποφασίζουμε να κάνουμε και εμείς έναν έλεγχο. Ταυτόχρονα. Και έχουμε διαπιστώσει πόσο σοβαρή και ποιοτική είναι η έλεγχη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι μονάχα να παρακολουθήσουμε τι κάνουν οι συναδελφοί μας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά να δούμε περί ποιων θεμάτων πρόκειται, ποια θέματα τους απασχολούν. Έχω τρία-τέσσερα παραδείγματα που είδα τέτοιοι συνοδευτικοί έλεγχοι που κρατούν τρεις-τέσσερις μέρες και που έγιναν δειγματοληπτικοί, έγιναν δειγματοληπτικά και που γίνονται στον τελευταίο δικαιούχο. Αυτό ήταν ενδιαφέρον για να γίνει και ένας έλεγχος από πλευράς Αυστριακού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για παράδειγμα, για το πρόγραμμα Leader ή για τα γεωργικά μέτρα. Κάναμε και εμείς έλεγχους. Έχουμε, για παράδειγμα, τώρα έναν έλεγχο για τις δημοσιονομικές διορθώσεις, που είναι σημαντικές και για την νομιμότητα και για την αξιοπιστία, για τη δήλωση αξιοπιστίας δηλαδή. Αποφασίσαμε να κάνουμε σχετικό έλεγχο και συντάσσουμε έκθεση. Συνολικά δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο χαίρει μεγάλου κύρους στην Αυστρία, αλλά και στο επίπεδο των επαφών έχουμε θαυμάσιες σχέσεις εμείς ως Αυστριακοί με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο που αντικατοπτρίζεται άλλωστε και στην συνεργασία μας σε πολλές ομάδες εργασίας. Μίλησα ήδη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Κύριε Μίλτερ, για σας, για το ποσοστό σφάλματος. 2% με ρωτήσατε είναι πολύ ή λίγο. Η ερώτηση σας είναι δύσκολη. Και βέβαια αυτήν κανονικά καλύτερα να την απαντήσει το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει και χρυσός κανόνας. Γνωρίζουμε ότι 2 έως 5% είναι λίγο πολύ ανεκτό σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα. Και εμείς στην ε, Αυστρία βάλαμε ένα κατόφλι. Με πρώτο κριτήριο, ποια είναι τα αντικείμενα που, που ελέγχουμε. Κυρίως μικρότερα πράγματα και εφόσον τα βγάλουμε αυτά απ' έξω, ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος στα ουσιαστικά. Για παράδειγμα, εάν διαπιστώσω ότι σε ένα έγγραφο δεν φέρει όλες τις υπογραφές ή αν διαπιστώσω ότι δεν έχει τηρηθεί μια διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού. Έχει διαφορετικό βάρος αυτό. Και εκεί αναλόγως πρέπει να κάνω και την ε, κριτική μου. Και βεβαίως πάντοτε υπό το πρίσμα του, της ανάλυσης κόστους ωφέλους. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάτι είναι υπερβολικό ή λιγότερο υπερβολικό. Και τώρα για την κοινή διαχείριση των πόρων. Προσπαθούμε πολλά να τα διαπιστώσουμε εκ των υστέρων. Να κάνουμε πρόσθετες δηλώσεις δηλαδή, για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Εγώ νομίζω όμως ότι πρέπει να πάμε στη ρίζα, εκεί όπου γίνονται οι πληρωμές, όπου γίνονται οι τελικές εγκρίσεις. Από εκεί πρέπει να αρχίσει ο έλεγχος. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξοικονομήσουμε και πολλούς πόρους. Δηλαδή ένας έλεγχος και καλός και όχι να προσπαθούμε βαθμιδών να κάνουμε όλο και περισσότερους ελέγχους που είναι και περισσότερο δαπανηροί. Τώρα, όλο και πρόσθετες δηλώσεις, οι οποίες επίσης πρέπει να ελεγχθούν μετά. Ίσως αποδίδουν μεγαλύτερη αξιοπιστία, αλλά νομίζω ότι και εδώ πρέπει κανείς να έχει υπόψη του το κριτήριο του κόστους και του ωφέλους. Εσείς τώρα με ρωτήσατε για τις δαπάνες και τα προγράμματα. Λέτε ότι το ελεγκτικό συνέδριο αντιμετωπίζει προβλήματα με την νομιμότητα των δαπανών. Και εγώ θα ρωτήσω για τη σκοπιμότητα. Οι ελεγκτές μπορούν να κάνουν και τα δύο. Έχουν την απαραίτητη παιδεία. Οι ερωτήσει άλλωστε είναι οι ίδιε. Μόνο τα συστήματα είναι διαφορετικά. Και καταλήγουν σε διαφορετικά αποτελέσματα ξαναλέω ότι δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα μείγμα. Στον έλεγχο της νομιμότητας, εφόσον ανακύψουν κάποια προβλήματα τα οποία έχουν σχέση και με τη σκοπιμότητα της δαπάνης, πρέπει να δώσουν αφορμή και για, μια, για έναν έξτρα έλεγχο. Έτσι νομίζω ότι μπορεί κανείς να συνεργαστεί καλύτερα και να είναι συμπλήρωση το ένα του άλλου. Για τον κύριο Έρενχάουζερ, τέσσερις ερωτήσεις μου έκανε. Αν είμαι φίλος του Μίχαελ Σπίντελεκερ. Απάντηση. Τον γνωρίζω από δύο συναντήσεις που είχαμε. Τη μία σε μία δημόσια εκδήλωση με 300 παρισταμένους όπου πέρασε σε ένα γύρο και μου έδωσε το χέρι του και με συνέστησαν ως ελεγκτή και αλλάξαμε λίγα λόγια τα οποία δεν θυμούμε καν, δεν είχαν καμία μεγάλη σημασία και άλλη μια φορά τον συνάντησα στο αεροδρόμιο στην Βιέννη με την σύζυγό του που ήταν τμήματάρχης στο δικό μου τμήμα και αυτός επέστρεφε από διαπραγματεύσεις στη Βόνη για την ε, βελτίωση του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Εκεί ο κ. Σπιντελέκερ είχε πάει να υποδεχτεί τη σύζυγό του στο αεροδρόμιο και πάλι εκεί του έδωσα το χέρι. Δεν έχουμε καμία ιδιαίτερη προσωπική φιλία ή επαφές και ούτε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή συμφέρον. Για μένα δεν τίθεται θέμα δηλαδή, ούτε και περαιτέρω ενδεχόμενα ε, επηρεασμού μου. Τώρα, αν η κυρία Σπίντε λέγεται θα συμμετάσχει στο προσωπικό μου γραφείο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, όπως θα είδατε και από τις απαντήσεις μου, έχω προετοιμαστεί πολύ εντατικά για την ε, σημερινή συνέντευξη. Και εφόσον όντως εγκαταλείψω το αξίωμά μου στο Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο για να έρθω εδώ, θα πρέπει να ολοκληρώσω κάποιε διαδικασίε. Έχω σπάσει το κεφάλι μου για όλα αυτά. Ωστόσο δεν έχω σπάσει το κεφάλι μου για το τι θα κάνω και ποιον θα αποκλείσω ενδεχομένω από το προσωπικό μου γραφείο στο μέλλον. Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν και περιφρόνηση και προ το ελεγκτικό συνέδριο και προ το κοινοβούλιο, εάν προαποφασίσω τα πράγματα αυτά. Γι' αυτό το λέω. Υπάρχει ένα αριθμό ε, υποψηφιότήτων που έρχονται και μου υποβάλλουν διάφοροι για να προσληφθούν, αλλά δεν έχω ακόμα απολύτως καμία ιδέα. Για την ακρόαση τώρα, για την ε, Επιτροπή του Αυστριακού Κοινοβουλίου. Χάρηκα όταν η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, που αποτελείται από συνασπισμό δύο κομμάτων, όταν διορίστηκε λοιπόν η κυβέρνηση αυτή, εγώ κατέθεσα την υποψηφιότητά μου για την θέση στο Ελληνικό Συνέδριο και ως γνωρίζετε στην Αυστρία απαιτείται η υποψηφιότητα αυτή που είναι απόφαση της αυστριακής κυβερνήσεως να εγκριθεί και από την Βουλή. Επιβεβαίωσε λοιπόν την υποψηφιότητά μου και το κοινοβουλευτικό επίπεδο και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα, κατά πόσον και αν στο παρελθόν έχουν γίνει ακροάσεις των υποψηφίων, αυτό δεν το ξέρω. Στην περίπτωσή μου πάντως δεν διεξήχθη ακρόαση. Και μια τέταρτη ερώτησή σας, κύριε Χάουζερ, δυστυχώς δεν διαβάζω τα γραμματά μου. Α, άλλοι υποψήφοι. Δεν γνωρίζω άλλον υποψήφιο. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος έχει υποβάλει υποψηφιότητα και δεν γνωρίζω εάν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο. Σας ευχαριστώ. Και τώρα μερικοί από τους συναδέλφους αρχίζουν να δυσφορούν γιατί θέλουν να συνεχίσουν τις ερωτήσει. Έχω ακόμα τον κύριο Ρούιμπιχ, τον κύριο Χατζημαρκάκη, τον κύριο Μίλντερ. Και κλείνω. Ο κύριος Ρούιμπιχ έχει το λόγο. Σύντομες ερωτήσεις για να έχουμε και σύντομες απαντήσει παρακαλώ. Κύριε Χέρεξ, σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω ιδιαίτερα για την παρουσία σας. Ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη. Είναι χαρακτηριστικό αυτό και αυτό νομίζω ότι ήδη είναι πολύ ε, καλό για τη σχέση μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριο κύριος Χατζημαρκάκης. Ναι, και εγώ θέλω να συμφωνήσω με τον Παύλο Ρούμπιχ. Μιλήσατε με μεγάλη εφράδια. Ήσασταν πολύ ε, καλά προετοιμασμένο, πολύ θετικό αυτό. Απλώ θέλω να ρωτήσω εάν η προκήρυξη τη θέση που γίνεται σε εσωτερικό επίπεδο στην Αυστρία και φαίνεται ότι ο τωρινός τώρα ε, εκπρόσωπος Αυστρίας στο ελεγκτικό συνέδριο διορίστηκε από την Αυστριακή κυβέρνηση. Αυτή λοιπόν η, η προκήρυξη, από ό,τι λένε οι αυστριακές εφημερίδες, ε, καθυστέρησαν εσκεμένα από τον αναπληρωτή καγκελόριο Σπέντλεκε, Κύριο Μίλτερ. Ίσως να μην άκουσα την απάντηση και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά ρώτησα εάν η Αυστρία μπορεί να έχει σε ομοσπονδιακό ή σε κατώτερο περιφερειακό επίπεδο ε, πιστοποίηση διαχείρισης. Ευχαριστώ και σας παρακαλώ να δώσετε απαντήσεις σε, στις πολύ συγκεκριμένε και σύντομες ερωτήσεις των συναδέλφων με τον ίδιο συγκεκριμένο και α, σαφή τρόπο και σύντομο. Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη τοποθέτηση, δεν χρειάζεται να σχολιάσω. Θα περάσω σε ερωτήσεις ε, για τον προκάτοχο δεν έχω ιδέα. Εγώ έχω υπόψη μου μόνο την προκήρυξη στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αυτό είναι το μέσο στο οποίο ανακοινώνονται οι προκηρύξεις, οι προκηρύξεις θέσεων και σε αυτό ανταποκρινόμενος κατάθεσα την υποψηφιότητά μου. Για τον κύριο Μίλτερ, εάν δεν, γι... δεν γίνονται αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους πιστοποίησης σε τοπικό, ούτε σε ομόσπονδο, ούτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Αυστρία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και ιδιαίτερα ευχαριστούμε για αυτή την εντατική ανταλλαγή απόψεων. Όπως είπαν και ο κύριο Ρίμπιχ και ο κύριος Χατζημαρκάκης ήταν πολύ καλά προετοιμασμένο δώσατε σαφεί απαντήσεις. Άλλο συνάδελφος δεν έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ θερμά. Και έτσι τώρα, και κλεισμένων των θυρών, συνεχίζουμε για τη συζήτηση. Παρακαλώ όσους ε, κυρίους και κυρίες ε, βρίσκονται εδώ και περιμένουν για το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη να αποχωρήσουν από την αίθουσα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Ah ja, okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης του υπαρχούν. Πέντε. Πριν όμως πούμε πάλι στην ε, ημερήσια διάταξη στο δημόσιο τμήμα. Θα ήθελα να ανακοινώσω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού εξέφρασε την υποστήριξή της και την εμπιστοσύνη στον κύριο Χέριξ κατά πλειοψηφία. Και έτσι περνώ στο επόμενο θέμα, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη με τον κύριο Γιάν Μιούλντερ. Έχουμε και τον κύριο Πίξιν εδώ. Καλώς ήρθατε. Ρωτώ τον εισηγητή εάν θέλει το λόγο ή θέλει να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο του λεπτικού συνεδρίου πρώτο, τον κύριο Πίξεν. Παρακαλώ λοιπόν να λάβετε το λόγο, κύριε Πίξεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να είμαι ειλικρινής δεν έχω να κάνω συγκεκριμένα σχόλια. Νομίζω ότι συνολικά Η έκθεση που μας προτείνει ο κ. Μούλντερ ευθυγραμμίστε σε μεγάλο βαθμό με τις παρατηρήσεις που είχαμε διατυπώσει στο συγκεκριμένο κεφάλι της ετήσιας μας έκθεσης και αν ο συνάδελφός σας, συζητητής κύριος Μούλντερ, ε, μάλλον και ο κύριος συζητητής σας ε, τονίζει τα σημεία που και εμείς είχαμε τονίσει. διεθνείς οργανώσεις ε, για και τα κονδύλια που δαπανώνται. Ήταν ένα σημαντικό ε, σημείο και διατυπώνει διάφορα επιχείρηματα ο κύριος Μούλντερ. Ίσως ένα πράγμα που μπορώ να αναφέρω εγώ είναι ότι το ποσοστό σφάλματος είναι υψηλότερο από αυτό που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Πάνω από το 3%. Πρέπει να γίνει λοιπόν δουλειά ε, για τη Europaid ε, αναφέρομαι εδώ και βέβαια και από το προσωπικό. Αυτά έχουμε να πούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο Ιαν Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, καθυσυχαστικό ήταν το σχόλιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στη δική μου έκθεση να πω πρώτα απ' όλα ότι η κατάσταση παραμένει κάπως περίεργη με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Είναι εκτός ε, του προπολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα το Κοινοβούλιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι. Η Κομισιόν είναι όμως αρμόδια για την εφαρμογή, ε, για την υλοποίηση των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Ε, εμείς ελέγχουμε την Επιτροπή, άρα στο εκ των υστέρων έχουμε κάποιο έλεγχο και στο κομμάτι αυτό εν γέννη. Να πω ότι είμαι θετικά διακείμενος ως προς το αποτέλεσμα, ως προς την υλοποίηση της δράσης από την Κομισιόν είναι γύρω στο 3%, 3,63% ή 3%. Τώρα το ακριβές ποσοστό μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι χαμηλότερο σε ό,τι αφορά ε, το ποσοστό εκτέλεσης του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Βλέπουμε βελτίωση κάθε χρόνο λοιπόν και νομίζω ότι αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Φυσικά τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο, εξού και διατυπώνω ορισμένα σχόλια, τα οποία ευθυγραμμίζονται και με τις υποδείξεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχω τις αμφιβολίες μου και εγώ για τη δημοσιονομική στήριξη, αλλά είναι πολιτική η απόφαση, εμείς πρέπει να ελέγχουμε τα πράγματα και κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο έλεγχος. Αν δίνεται λοιπόν δημοσιονομική ενίσχυση, δημοσιονομική στήριξη, αυτό αποτελεί ε, μια σταθερή μας ε, μέρημνα. Ε, δεν νομίζουμε ότι είναι ιδεώδης η κατάσταση προς το παρόν τουλάχιστον. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Κονκό και την Αιτή. συμφωνώ με τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τώρα, συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ κτλ. Θα υπενθυμίσω κάτι που έχω πει σε πολλέ εκθέσεις κατά το παρελθόν. Ότι αν συνεργαστούμε με τέτοιου διεθνείς οργανισμούς όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, θα πρέπει να δούμε ότι το 95%, 90 με 95% ε, το καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρόγραμμα μιλάμε του ΟΗΕ. Και όταν πάει κανείς επί τόπου βλέπει σαν να είναι χρηματοδοτούμε 100% από τον ΟΗΕ και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό. Επίσης, τι είναι μια πραγματική μη κυβερνητική οργάνωση. Αν κάποιο συνεργάζεται με μια μη κυβερνητική οργάνωση θα πρέπει και η ίδια να συνεισφέρει. Επιτόπου συχνά διαπίστωσα ότι είναι ανύπαρκτη η συνεισφορά της ΜΚΟ. Και αν υπάρχει εισφορά, υπάρχει από την εθνική κυβέρνηση. Και αυτό νομίζω ότι ε, είναι σαν κοροϊδία για την ύπαρξη αυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης, αφού η κυβέρνηση χρηματοδοτεί. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και σε ό,τι αφορά την ε, ε, χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Τέλος, το μηχανισμός επενδύσεων είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο, συγκρίσουμε αυτό που ζητούμε να έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ένα Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο δηλαδή μιλώ, αλλά αυτός ο μηχανισμός επενδύσεων, investment facility, θα ήταν καλό ε, επειδή έχετε διάφορες χρηματοδοτήσεις, να ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης. Γιατί μέχρι στιγμής είναι μια κάπως άμορφη μάζα και δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού προέρχονται τα χρήματα και πώς ε, δαπανούνται. Αυτά είχα να πω για τη δική μου έκθεση κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. σε ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή κύριο Γιάν Μούλντερ και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Γενικός Γραμματέας Ντιμέλο, τον οποίο θέλω να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Σας παρακαλώ να μας ε, μιλήσετε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι τιμή που βρίσκομαι ενώπιον σας από τότε που ανέλαβα την Γενική Διεύθυνση της λεγόμενης Europe Aid. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι βουλευτές, ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε την έκθεση του κυρίου Μιούλντερ, πρώην συναδέλφου στην DG ε, Αναπτυξιακής Βοήθειας. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την ισορροπημένη αυτή και ουδέτερη αντικειμενική έκθεση. Έχουμε αρκετούς τομείς διαχείρισης του EDF με ποσοστό μειούμενο από το 5,1% στο 3% εφέτος. Αναγνωρίζει επίσης ο εισηγητής ότι ε, έχουμε στην ανάπτυξη πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε ε, δυσμενείς συνθήκες. Πολλοί είναι οι τομεί που καταγράφει και ο εισηγητή, στου οποίου θα πρέπει και εμεί να καταβάλουμε περισσότερε προσπάθειε. Θα ε, μελετήσουμε προσεκτικά αυτέ τι συστάσει, όπω άλλωστε έχουμε ήδη ξεκινήσει και θα τι λάβουμε και στο μέλλον υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο κύριο Μιούλτζερ και όλοι οι συναδελφοί του στην Επιτροπή σα, ξέρω ότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με το 3% ποσοστό σφάλματος που καταγράφεται από το ελεγκτικό συνέδριο. Ωστόσο, πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και επιβεβαιώνω τη βούλησή μας να προχωρήσουμε για περαιτέρω μείωση του λάθους. Το υπόλοιπο αυτό ποσοστό σφάλματος που έχει αναλύσει η ΔΕΦΚΟ μαζί με το ελεκτικό συνέδριο μας έχει προσφέρει και πολύτιμες πληροφορίες και μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τους πιο σημαντικούς ε, ε λόγους των σφαλμάτων με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια τροποποίηση στα συστήματά μας από το Σεπτέμβριο του 2013 που πιστεύουμε θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του ε, ποσοστού σφάλματος ώσπου να φτάσουμε και στο μηδαμινό σφάλμα στο ETF. Εδώ λοιπόν από το 2012 έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη μεταρρύθμιση της προσέγγισης μας για το EDF η νέα πολιτική έχει πλέον τεθεί πλήρως σε εφαρμογή το τελευταίο δεκάμινο. Ε, βλέπουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ε, σημειώνουμε ότι το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου ε, καταγράφεται στα θεωρητικά σχόλια της εκθέσεως. Σημειώνεται επίσης ότι έχουμε ένα υψηλού επίπεδου στρατηγική, στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου που έχει θεσπιστεί για την κάθε χώρα που ε, λαμβάνει χρηματοοικονομική υποστήριξη. Συνεχίζουμε λοιπόν τη δουλειά μας με το πλαίσιο αυτό διαχείρισης κινδύνου και περιμένω να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε και περαιτέρω αποτελέσματα στην Επιτροπή σας σύντομα. Απαιτείται, λέει η έκθεση, πιο αυστηροί όροι να εισαχθούν για την ε, επιλογή των δικαιούχων και την εκτέλεση των έργων αλλά και σε άλλε περιπτώσει για ορισμένε χώρες, δεδομένη μιας ιδιαίτερη πολιτική κατάσταση να περιοριστεί ή να είναι λιγότερο αυστηρή η όρη. Πιστεύω ότι μπορεί, αν είμαστε υπερβολικά αυστηροί, να ειναι λιγοτερο αυστηρη πιστευω οτι μπορει αν ειμαστε υπερβολικα αυστηροι να τεθει σε κίνδυνο όλο το εγχείρημα και η προσέγγιση μα. Θα πρέπει αυτέ οι καταστάσει δηλαδή να αξιολογούνται με όρου που δεν εξαντλούνται στου ε, αποκλειστικούς όρους για την ε, εκτέλεση των προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Γενικό Διευθυντή, κύριο Ντιμέλο. Και ακούμε τώρα τους συναδέλφους. Αρχίζει η συζήτηση στην Επιτροπή μας με την Ίγκια Κρέσλε πρώτα. Ευχαριστώ. Πολύ χαίρομαι κύριε Ντιμέλο που είστε εδώ και συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Γενικό Διευθυντή. Θα ήθελα ξεκινώντας να πω ότι τα ζητήματα που συζήτησε ο εισηγητής ε, με τη μη κυβερνητική οργάνωση έχουν μεγάλη σημασία. Είχα συμμετάσχει και εγώ σε μια ομάδα. Είδαμε ότι 1305 μη κυβερνητικέ οργανώσει αναλαμβάνουν δράση χρηματοδοτούμενες με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο χώρο του Europe Aid και του ECO. Είναι περίπου οι μισές οι κυβερνητικές οργανώσεις. Πολλά από τα κονδύλια πάνε μέσω της χρηματοοικονομικής υποστήριξης και βέβαια το ερώτημά μου είναι καταρχάς τα υπόλοιπα κονδύλια που πάνε. Άρα λοιπόν θα ήθελα να δω τα, τον έλεγχο καταρχάς των κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και το πολιτικό αποτέλεσμα, το political result. Τι δίνει. Ε, υλοποιούν τη δική μας πολιτική αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ή μήπως κάποιο δικό τους ε, θεματολόγιο, γιατί έχουμε κάποιες ε, επιφυλάξεις σε αυτό το θέμα. Επίσης, ε, προσπαθήσαμε να μελετήσουμε έγγραφα, ώστε να τον περισσότερα, και θα ήταν καλό να δούμε ένα συγκεκριμένο έγγραφο για την EMG, που να αποδεικνύει ότι είναι μια διεθνής, διεθνούς εμβέλειας οργάνωση με το ε, Διευθυντικό Συμβούλιο, το Steering Committee. Δεν βρήκαμε μας τέτοιο έγγραφο και θα θέλαμε να μας το εξασφαλίσετε. Μας λυπεί το γεγονός πάντως ακόμη ότι η μη κυβερνητική οργάνωση EMG φαίνεται να μπορεί να αποκομίσει κέρδος. Πράγμα το οποίο καταρχήν ίσως να μην είναι παράλογο. Διαπιστώνω πάντως ότι ο επικεφαλής, ο πρόεδρος της CMG είναι και ο ιδρυτής της. Ύστερα από 35 χρόνια που δραστηριοποιείται αυτή η οργάνωση έχει μείνει στην ίδια θέση. Άρα είμαι υποχρεωμένη να σας ρωτήσω δεν υπάρχει κάποια σύμβαση. Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος να είναι πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει έχει ιδρύσει μια επιχείρηση ιδιωτική την οποία ο ίδιος εξακολουθεί να ε, δεν είναι τότε κάτι άλλο από μη κυβερνητική οργάνωση αυτή η EMG. Και από την άλλη ξέρουμε ότι κάνει πολύ σημαντική δουλειά. Χαιρόμαστε που υπάρχει αυτή η οργάνωση. Αλλά είναι μια επιχείρηση όπως κάθε άλλη. Και αν είναι μια κοινή οργάνωση όπως κάθε άλλη, γιατί έχει πρακτική εδώ και δεκαετίες που δεν ταιριάζει σε μια επιχείρηση όπως κάθε άλλη, δηλαδή χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το υλικό που χρειάζεται να λάβουμε είναι η μη άλλο αρκετό, ε, είναι απαραίτητο, αν όχι, αλλά όχι επαρκές. Και δεν ήθελα έστω και διμερώς να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Δεν Θέλει κανείς άλλο το λόγο, ο Μπέρμαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. σε ό,τι αφορά το ρόλο της δημοσιονομικής ενίσχυσης και των ΜΚΟ, φυσικά και μπορούμε να το συστήσουμε διαμακρών, θα ήταν καλό ίσως να δούμε και τις προκηρύξεις διαγωνισμών όπου προσπαθούν οι ΜΚΟ να εκπληρούν ε, τα κριτήρια και τις ε, υποθέσεις της Κομισιόν που είναι πολύ υψηλές και πολλές φορές παραπονούνται οι ΜΚΟ για τη δυσκολία όλων αυτών των όρων που πρέπει να εκπληρώνουν. Ε, είναι σαφής βέβαια οι προϋποθέσεις και οι όροι και σίγουρα είναι σημαντικό να γίνεται ένας έλεγχος ενδελεχής και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά δεν θα ήταν τάση δική μου να είμαστε καχύποπτη να είναι αυτή η πρώτη μας αντίδραση απέναντι στις ΜΚΟ, γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα τα σχέδια και οι στόχοι των ε, προγραμμάτων μέσω των προκηρύξεων διαγωνισμών, που ναι μεν έχουν δικό τους όραμα πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, Χριστιανικέ μη και πολλά και διάφορες μπορεί να είναι αυτέ οι μη αλλά όταν είναι πολύ συγκεκριμένοι οι όροι που πρέπει να ε, εφαρμόζουν δεν έχουν ε, περιθώρια. Επίσης είχαμε συζητήσεις ε, με το ελεκτικό συνέδριο και νομίζω ότι ίσω θα ήταν καλό να υπάρχει μεγαλύτερη ανταλλαγή μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και Κομισιών σε ό,τι αφορά τον έλεγχο πολιτικών για τις οποίες ίσως ε, το Ελεγκτικό Συνέδριο ε, κάπως δυσκολεύεται να ε, αποκρυπτογραφήσει. Και εμείς, ξέρετε, πολλές φορές ζητάμε δείκτες, δείκτες ξεκάθαρους και μετρήσιμους, για να διευκολυνθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων και για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εμείς διατυπώνουμε με την νομοθεσία μας. Νομίζω ότι η Κομισιόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανάγκη να έχουν μεγαλύτερη συνεργασία και για τομείς που ίσως να είναι όχι τόσο εύκολο να μετρηθούν. Εκεί λοιπόν πιστεύω ότι θα ήταν καλό να συνεργάζεστε περισσότερο Κομισιόν και Ελεγκτικό Συνέδριο για να μην υπάρχουν αυτές οι εντάσεις και για να μην υπάρχει και αυτή η έλλειψη συνεννόησης και κατανόησης. Το είδαμε πριν από κάποιους μήνες ότι υπάρχει αυτό το αίτημα από πλευρά Ελληνικού Συνεδρίου. Δεν ξέρω, έγινε κάτι, δηλαδή εισακούστηκε το αίτημά του για μεγαλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή μεταξύ Κομισιών Ελεκτρικού Συνεδρίου. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Άλλο συνάδελφο που θέλει το λόγο. Παόλο Ριουμπίκ και μετά η κυρία Κρέσλα. Ευχαριστώ πολύ. Η χρηματοδότηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης με ενδιαφέρει εμένα. Δηλαδή, εάν μεταφέρονται κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη κυβερνητικές οργάνωσεις και καταλήγουν σε φορολογικούς παραδείσους ή σε εταιρείες offshore. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τέτοια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και η Ίγκε Γκρέσλε. Περιμένει. Ναι, θα ήθελα να πω στον κύριο Μπέρμαν ότι δεν είναι όλες οι NGO μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες παίρνουν την, αφρό, την και κάποιες άλλες ε, δεν είναι πάντα στην ίδια θέση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν καλό να μας πει ο Γενικός Διευθυντής τι είδους χρηματοδότηση παίρνουν οι μεγαλύτερες μη κυβερνητικέ οργανώσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Ανάπτυξης. Και ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Τώρα θα ακούσουμε από την Επιτροπή, κύριε Γενική Διευθυντά, για την απάντηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τον βουλευτές για τις ερωτήσεις σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω στο δυνατόν πληρέστερα. Πρώτα απ' όλα για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εμείς θεωρούμε στην Κομισιόν ότι μη κυβερνητικέ οργανώσει, ιδίω στον αναπτυξιακό τομέα, έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και συμβάλλουν στι αναπτυξιακέ πολιτικέ, όχι μόνο με τη συμμετοχή του στη διαχείριση των διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων, αλλά και με την συμμετοχή μέσω της κοινωνίας των πολιτών, που η συνεισφορά της είναι πολύ χρήσιμη. Επομένως, έχουμε προβεί σε θετική αξιολόγηση της κοινή δουλειά που κάνουμε μαζί με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ό,τι αφορά τώρα τη χρηματοδότηση, κατά την υπογραφή μια σύμβασης με μια ΜΚΟ, πάντοτε αναφέρεται το ποσοστό του έργου, του σχεδίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ή το ΕΤΕ, το, Ευρωπαϊκό Ταμείο, ε, το ΕΤΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και, γίνει, και κάνουμε τους λογαριασμούς, ε, την εκαθάριση, βλέπουμε ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης που αντιστοιχούσε στη ΜΚΟ έχει καλυφθεί. Τι συμβαίνει όμως ενίοτε. Η πηγή χρηματοδότηση δεν είναι πάντοτε ίδια με αυτή που είχε αναγγελθεί στην αρχή. Σύνηθε το φαινόμενο λόγω της φύσης των ΜΚΟ και των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης. Ενδέχεται δηλαδή να έχουν ε, ανακοινώσει κατά την υπογραφή της μας μια άλλη πηγή χρηματοδότησης και όταν στο τέλος ελέγχουμε κατά πόσον ε, δόθηκαν τα χρήματα αυτά, ε, βλέπουμε κάποιες φορές μια διαφορετική πηγή χρηματοδότησης. Αυτό όμως δεν αμφισβητεί ε, τη συμμετοχή. Το θέμα είναι ότι παραμένει ίδιο το δικό μας ποσοστό συμμετοχής, το δικό μας ποσοστό συγχρηματοδότησης. Αυτό νομίζω ότι είναι σύνηθε σε τέτοιες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, γιατί λαμβάνουν χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές και επαναλαμβάνω ένα φαινόμενο που μπορεί να συμβεί. Κατά την άποψή μας αυτό όμως δεν αμφισβητεί την ε, κανονικότητα της συγχρηματοδότησης από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό βέβαια είναι να επιτευχθούν τα αποτελέσματα και να τηρηθούν οι κανόνες. Σε ό,τι αφορά την IMG, νομίζω ότι είχαμε δώσει μια πάρα πολύ εντελεχή απάντηση ε, στα ερωτήματα που έθεσε η δική σας επιτροπή και όχι μόνο μία φορά, την τελευταία φορά πριν από ένα μήνα. Σε 170 ερωτήσεις ε, έχουμε απαντήσει ε, για το IMG, τη Διεθνή Διαχειριστική Ομάδα. 70 σελίδες ήταν οι απαντήσεις μας. Τι μπορώ να σας πω σήμερα λοιπόν. Μπορώ να σας πω ότι η IMG, η Διεθνής Διαχειριστική Ομάδα, συγκροτήθηκε με συμμετοχή πολλών κρατών μέλων, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι συμμετέχουσες χώρες. Αυτή η διαχειριστική ομάδα εργάζεται ή συνεργάζεται και με πολλά άλλα κρατημέλη, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Κροατία. Εργάζεται και με, τρίτα, με τρίτους, ε, όπως Νορβηγία, Ελβετία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Πολλές λοιπόν αναπτυξιακές, πολλοί αναπτυξιακοί φορείς και πολλές χώρες και τρίτες χώρες συνεργάζονται με αυτή την ομάδα και εξ όσων γνωρίζουμε δεν αποκομίζουν κάποιο κέρδος, ε, έχουν αποτελέσματα τα οποία μεταφέρονται στη νέα διαχειριστική χρήση. Δεν κατανέμονται, δεν ε, πηγαίνουν σε κανέναν μεταφέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος. Βέβαια είναι ένα θέμα ότι έχουν πλέον ε, εμπειρία, τεχνική, τεχνογνωσία, ώστε σε διαφόρους τομείς, ε, επειδή έχουν ακριβώς αυτή την εμπειρία, δεν μπορεί κανείς να τους παρακάμψει και να στραφεί αλλού. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, διακόπτουμε τις συμβάσεις αυτές και περνάμε στην κανονική διαδικασία ε, προκήρυξης διαγωνισμού. Στην περίπτωση του προγράμματος ε, που αφορούσε την Παλαιστινιακή Αρχή, αποφασίσαμε να διακόψουμε την σύμβαση με την IMG και τον προηγούμενο Νοέμβριο προκηρύξαμε έναν διαγωνισμό. Περάσαμε δηλαδή στις κανονικές ε, περιστάσεις, κανονικές συνθήκες αλλά σε χώρες που βρίσκονται ε, σε περίοδο μετά από ε, εμπόλεμη σύραξη και εμείς και άλλοι εταίροι ε, προσφεύγουμε στην ομάδα αυτή λόγω της εμπειρίας που έχει συγκεντρώσει στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά το θέμα των σαφών δικτών που σχετίζονται και με τα αποτελέσματα των πολιτικών, εδώ υπάρχει μια μια διπλή διάσταση. Η μία διάσταση βέβαια είναι ότι όταν ορίζονται τα προγράμματα, θέλουν όλοι πώς να το πω, να είναι πάρα πολύ θετική και φιλόδοξη σε σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ιδίω δε οι πολιτικοί πάντοτε θέλουν να είναι πολύ φιλόδοξοι. Πολύ συχνά κατά την κατάρτιση και την ανάπτυξη επιτόπου του προγράμματος είναι δύσκολο ή, δεν, ε, ή αδύνατο να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα, αυτοί οι στόχοι. Άρα πρέπει να ορίζονται ε, στόχοι που να είναι ρεαλιστικοί. Εξού και ε, εμεί εισαγάγαμε μια νέα προσέγγιση για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Results Framework Approach. Αυτή θα είναι η νέα προσέγγιση που θα ενταχθεί σε όλα τα ενδεικτικά προγράμματα του 11ου Γιατί το κάνουμε τώρα. Θα δείτε, θα δείτε σύντομα ε, ότι στα ενδεικτικά προγράμματα θα έχουμε την ίδια δέσμη δικτών, οπότε είναι δυνατόν να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων στις διαφορετικές χώρες. Αναθεωρούμε λοιπόν ε, τους δείκτες μας, έχουμε πλέον ε, ορίσει ορισμένους δείκτες που θα ισχύουν παντού, που είναι μετρήσιμοι, γνωρίζουμε ότι θα μπορούμε, ε, γιατί έχουμε τα στατιστικά δεδομένα να τους καταρτήσουμε, θα έχουμε και αυτά τα stress test, αυτές τις δοκιμές αντοχής και επομένως έχουμε την πεποίθηση ότι και τη βεβαιότητα θα έλεγα ότι μπορούν να λειτουργήσουν οι δείκτες αυτοί για να γνωρίζουμε καλύτερα ποια είναι και ποια θα είναι τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και για τους σκοπούς της δικής μας διαχείρισης αλλά και για τους σκοπούς της ε, λογοδοσίας ώστε να μπορεί και το Ελεκτικό Συνέδριο και το Κοινοβούλιο να ελέγξουν τους δείκτες και τα αποτελέσματα. Και είπα, οι δείκτες θα είναι οι ίδιοι στα διάφορα προγράμματα. Ελπίζω λοιπόν με αυτή την προσέγγιση να είμαστε σε θέση καλύτερα να ορίσουμε και να ελέγξουμε και να επανελέγξουμε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Yeah, thank you very much. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Πίνξτιν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αν θέλετε να απαντήσετε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για σημαντική συζήτηση. Έχω ορισμένα σχόλια. Πρώτο, ποιες είναι οι τάσεις τα τελευταία χρόνια διαμορφώνονται οι τάσεις ώστε στα μέσα της προθεσμίας περισσότερα χρήματα έχουν δαπανηθεί για στήριξη του προϋπολογισμού με των οργανισμών του ΟΗΕ και περισσότερα χρήματα έχουν ταπανηθεί από μη κρατικέ οργανώσεις. Πρόκειται για μια τάση που περιπλέκει τους ελέγχους. Δεύτερο σχόλιο. Εάν δαπανώνται περισσότερα χρήματα με έμεσο τρόπο, όπως εξήγησα στο πρώτο μου σχόλιο, γίνεται πιο σημαντικό να διεξάγονται μετρήσεις των αποτελεσμάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν δείκτες, χρειαζόμαστε τα αποτελέσματα να συγκρίνονται μεταξύ των χωρών και τα αποτελέσματα να είναι καθαρά μετρήσιμα. Τρίτο σχόλιο, η αρεσιμότητα. Θέμα ευαίσθητο, εάν όμως είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε οι χώρες μέλη αποφασίσουν να δαπανούν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάση αιρεσιμότητας, δεν μπορεί να αναμένει κανείς από το ελεγκτικό συνέδριο να μην ελέγχει τους όρους, την αρεσιμότητα δηλαδή. Βεβαίω γνωρίζουμε ότι πρέπει να εξευρεθεί η ορθή σχέση ισορροπία ανάμεσα στους όρους της αρεσιμότητας δηλαδή από τη μια μεριά και σε κάποια ρεαλιστική σχέση από την άλλη. Όμως εάν γράφεται στα έγγραφα της Κομισιόν ότι περιλαμβάνονται όροι, βεβαίως τότε εξετάζουμε τους όρους και ελέγχουμε δαπανήθηκαν τα χρήματα με σεβασμό των όρων που επιβάλλουν τα έγγραφα, οι συνθήκες κλπ. Και αυτό θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε να πράττουμε, ακόμα και αν ορισμένες φορές θα πρέπει να εμφανιστούμε ρεαλιστές απέναντι σε εύθραυστες χώρες κτλ. Αλλά πιστεύουμε και πιστεύω και εγώ προσωπικά ότι οφείλουμε να εξετάζουμε, όπως είπα, τους όρους. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πάντοτε και τα δύο. Και ήταν πίτα ολόκληρη και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή ως κοινοβούλιο να λέτε από μια μεριά ότι θέλουμε σεβασμό της δημοκρατικής νομιμότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λοιπά στις χώρες όπου θα πανούμε τα χρήματά μας και από την άλλη μεριά να λέμε α ναι αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές διότι και λοιπά η συζήτηση θα πρέπει να είναι σαφής και ξεκάθαρη. Το συνέδριο εξετάζει τα έγγραφα, τα γεγονότα, τους όρους και μετά το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα πει τι είναι αποδεκτό για τα όργανα αυτά και τι όχι. Εάν το Κοινοβούλιο πει κάποτε ότι προς χάρη κάποιας ρεαλιστικής λύσεως σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου ή ευάλωτες χώρες κλπ. θα πρέπει να τα εξετάσουμε τα πράγματα, τους όρους δηλαδή, την εφαρμογή των όρων κάπως διαφορετικά, έστω. Αλλά πάντως εμείς πιστεύουμε ότι η συζήτηση τουλάχιστον πρέπει να είναι πολύ σαφής. Αυτά ήταν τα τρία σχόλια που ήθελα να κάνω από τη δική μου πλευρά. Επαναλαμβάνω ότι το έγγραφο είναι ενδιαφέρον, καθώς και η συζήτηση. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίξτεν. Κύριε Μίλτερ, είστε ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. να το ξεχάσω. Έπρεπε όμως στην αρχή να έχω αναφέρει ότι είμαι πρώην ε, της τη ε, Γενική διεύθυνση για την Αναπτυξιακή Βοήθεια. Είχαμε πριν από 30-40 χρόνια με τον κύριο Ντιμέλο αυτά τα καθήκοντα αναλάβει. Εγώ πιο νωρί ίσω. Εγώ το 94 αποχώρησα πριν από 20 χρόνια. Ο κύριο Ντιμέλο ήταν σοφό και έμεινε. Και κατάφερε αυτό που όλοι περιμέναν ότι θα κατάφερνε να γίνει γενικό διευθυντή. Άρα σοφά επέλεξε να παραμείνει στη Γενική Διεύθυνση για την Ανατολική Βοήθεια. Για τη συζήτησή μα τώρα, για το θέμα των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ε, ο προβληματισμό δεν είναι καινούριο. Ήδη το 2004 σε ψήφισμα το ζητούσε το Κοινοβούλιο από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συντάξει μία ειδική έκθεση για την Ανατολική βοήθεια σε διεθνεί οργανώσει και με κυβερνητικέ οργανώσει. Δύο εκθέσει που ε, δύο χρόνια αργότερα μόλι δημοσιεύτηκαν ε, η έκθεση που αφορούσε τι διεθνεί οργανώσει ήταν πολύ καλή. Η έκθεση για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει απογοητευτική, κυρίω διότι για μένα τουλάχιστον δεν κατέστη ποτέ σαφέ τι είναι μη κυβερνητική οργάνωση, πώ ορίζεται. Εάν λοιπόν μια μη κυβερνητική οργάνωση οργα... ε, ε αναγνωρίζεται ω τέτοια από κράτο μέλο ή από κράτη-μέλη, μα είπαν από, από την Γενική Διεύθυνση, ε, από το ελεκτικό συνέδριο, άρα είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, διότι δεν ξέρουμε με τι κριτήρια να γνωρίζει ω μη κυβερνητική οργάνωση ένα κράτο μέλο μία οργάνωση. Λοιπόν, εγώ μπορεί να έχω επαφέ πολλέ με μη κυβερνητικέ οργανώσει, συζητώ και γνωρίζω πολλά μέλη του και εκπροσώπου του, αλλά χωρί να αμφιβάλλω ότι πολλέ από αυτέ κάνουν πολύ καλή δουλειά ω μη κυβερνητικέ οργανώσει, είμαι βέβαιο ότι δεν είναι όλε έτσι. Εξού και οι ανησυχίες και επιφυλάξεις μου. Γιατί μιλώ σε μια μη κυβερνητική οργάνωση, με μια κυβερνητική οργάνωση παραδείγματα για διάφορα θέματα μη, ε, ανθρωπινών δικαιωμάτων και όταν έρχεται η ώρα να ρωτήσω από πού προέρχεται η χρηματοδότησή τους, η απάντηση που λαμβάνω είναι μα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά. Και όταν ρωτάω, εντάξει, πλην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλο κανεί σα χρηματοδοτεί, Παίρνω την απάντηση συνήθω όχι. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μα χρηματοδοτεί. Πράγμα το οποίο κατά την έποψή μου δεν είναι ο τρόπο λειτουργία μια μη κυβερνητική οργάνωση. Μια κυβερνητική οργάνωση για διάφορου λόγου ξεκινάει από κάποιου ανθρώπου που θέλουν να προωθήσουν έναν σκοπό, έχουν τον ενθουσιασμό του, την προσωπική του εργασία και όλα αυτά και συμπληρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδότηση. Αν ήταν να χρηματοδοτεί 100% ε, μια οργάνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αναλάβει να αναθέσει μάλλον σε κάποιον ε, αντισυμβαλόμενο. Και ναι, μπορεί κάποιοι να κάνουν καλή δουλειά όπως είπα, αλλά από τα στοιχεία που έχουμε το 2004 είχαμε 1,3 δις, γιατί θυμάμαι πολύ καλά αυτά τα στοιχεία τότε που ήμουν ακόμα πιο ε, Ενεργώ σε αυτά τα θέματα. Ε, πολύ μικρό ποσοστό πήγαινε μέσω προκηρύξεων στον ε, πλειοδότη. Η δε συντριπτική πλειονότητα των ποσών αυτών, το 70 περίπου πήγαινε απευθείας σε 100% χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και πολλές φορές ε, έχουν και επιδότηση ιδιαίτερη, γιατί βέβαια ξέρουν τα κόλπα και τα γρανάζια. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το ηλεκτρικό συνέδριο και με έκπληξη ακούω ότι σε σχέση με το 2004, το 2014 ο προϋπολογισμός αυτός έχει διπλασιαστεί μέσα 10 χρόνια. Η κυρία Γκρέσλε χωρίς μικρόφωνο. Έστω, σε αυτό το τομέα μόνο, αλλά πάντως βλέπω ότι έχει διπλασιαστεί, είναι σημαντική αύξηση και αποτελεί ασφαλώς ένα λόγο επιπλέον να μελετήσει πιο προσεκτικά το ελεκτικό συνέδριο αυτό το πράγμα. Για τα υπόλοιπα δεν έχω άλλα σχόλια. Θέλω απλώ να υπογραμμίσω ότι απαιτείται μια ενδελεχής εξέταση του Ευρωπαϊκού Μέσου Επενδύσεων για την Αφρική. Πάλι έχουμε να κάνουμε 2 δισεκατομμύρια, πολύ σημαντικό ποσό και δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς λειτουργεί η διάθεση των κονδυλίων, τι, τι μηχανισμός υπάρχει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τώρα θα κάνουμε ένα σύντομο γύρο συζητήσεως ο κύριος Μπέρμαν. Κύριε Πρόεδρε, λίγο ε, ηρωνικό μου φαίνεται που ο αγαπητός συνάδελφος ε, Γιάν Μούλντερ δεν είναι ικανοποιημένος με την ιδέα του ότι ενίοτε ε, 100% κρατική είναι η χρηματοδότηση που παίρνει μια ΜΚΟ. Τι θέλετε, θέλετε να τους, κάνε, ε, τους κάνουμε μια κυβέρνηση, ε, να τους κάνουμε κρατικούς υπαλλήλους, νομίζω θέλουμε μια μικρή κυβέρνηση. Δεύτερον, πολύ πολιτική, περισσότεροι πολιτική, θα ήταν πάρα πολύ ε, ικανοποιημένοι αν οι ίδιοι είχαν ποσοστό σφάλματος στις τάξεις του 3%. Κανείς δεν υπολογίζει το δικό μου ποσοστό σφάλματος, λέει ο κύριος Μιλντερ. Ε, ε, ε, κύριε Κρέσλε. Ναι, αλλά αν ήταν τόσο χαμηλέ οι προϋποθέσεις θα Αν ήταν τόσο αυστηρέ προποθέσει και στο θέμα αυτό, θα είχαμε ποσοστό σφάλματος κάτω από το 2% μηδαμινό. Αυτό που με ενοχλεί πάντω σε μένα είναι ότι φαίνεται να ολοκληρώνουμε μια συζήτηση μόνο με συμπέρασμα τι καλά που τα πάμε. Δεν αρκεί αυτό. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, πρέπει να ξαναμελετήσετε όλη αυτή την πληθώρα των έργων και των προγραμμάτων και να προσπαθήσετε να οργανώσετε καλύτερα την ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μην ξεχνάμε ότι το, το κτίριο αυτό του Φαν Ρόμποϊ πίσω στη γωνία κάνει 300 εκατομμύρια ευρώ. Κοστίζει 300 εκατομμύρια ευρώ ένα μόνο κτίριο. Ίσως καλό θα ήταν ε, ε, να σκεφτούμε αυτά τα δύο δις που προβλέπονται ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση πόσο χρήσιμα θα μπορούσαν να ήταν και πόσα πολλά έργα θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν. Μήπως αντί να έχουμε κατακαιρματισμένα μικρά έργα θα ήταν πιο σκόπιμο να, τα, να ενοποιήσουμε τα κονδύλια και τα προγράμματα, να έχουμε έργα βάσης ανάλογα και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αυτό είναι ένα θέμα επιλογής. Πρέπει να δούμε, θα την ενοποιήσουμε, τη βοήθεια την ε, ομαδοποιήσουμε καλύτερα ή θα συνεχίσουμε όπως τώρα. Μπήκαμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχουμε συζητήσει παλαιότερα και με τον κύριο Πίμπαλξ, επίτροπο. Και είχα ρωτήσει εγώ τότε εάν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι σε μη κυβερνητικέ ή μη κρατικές οργανώσεις και σε ορισμένες προβληματικές περιοχές να μην καταλήξουν τα χρήματα σε λάθος χέρια. Γιατί σε ορισμένες περιοχές του Πακιστάν, για παράδειγμα, είχαμε ένα πρόβλημα με ένα σημαντικό ποσό που πέρασε από την Αίγυπτο. Και πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων δεν καταλήγουν ενδεχομένω και σε έμεση χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Σε χώρες που βρίσκονται σε σημαντικές κρίσεις ή που έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια να μπορούν να διατεθούν κονδύλια με τρόπο γρήγορο και όχι γραφειοκρατικό εάν υπάρχει θεομηνία παλιροϊκό κύμα, ε, σεισμός και ούτω καθεξής, να είναι δυνατό και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία βλέπει λογαριασμούς. Εκεί όμως όπου διατίθεται βοήθεια μακροπρόθεσμα σε χώρες πρέπει να εξετάζονται οι τελικοί δικαιούχοι. Θυμίζω και την έκθεση Μπέρμαν για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις βοήθειες στη Λωρίδα της Γάζας. Σημαντικό πολιτικά θέμα. Κύριε Γενική Διευθυντά, ίσως μπορείτε να πείτε λίγα λόγια τώρα για τις ερωτήσεις που μόλις ακούσατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα θέματα που θέσατε είναι δύσκολα βέβαια και πολύ ε, σημαντικά πολιτικά, με σημαντική πολιτική διάσταση βέβαια Διαρκώς καλούμεθα να λαμβάνουμε, να λαμβάνουμε αποφάσεις. Εάν είναι δηλαδή απαραίτητο να αναλυφθούν κάποιοι κίνδυνοι, είτε στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης, για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους σε δύσκολες καταστάσεις, το οποίο συνήθως πράττουμε, ή εάν θα πρέπει να μην κάνουμε κάτι για να είμαστε ασφαλείς. η Επιτροπή, αλλά νομίζω και το Κοινοβούλιο, πιστεύω, είναι υπέρ της παρεμβάσεως σε τέτοιες περιπτώσεις και της ανάληψης των σχετικών κινδύνων σε χώρες όπου σημειώνονται συγκρούσεις ή σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, θεομηνίες και ούτω καθεξής, όπου συχνά είναι πάρα πολύ δυσχερές να παρακολουθηθούν, μάλλον συγγνώμη, να τηρηθούν όλοι οι σχετικοί κανόνες και έλεγχοι που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Μερικές φορές έχουμε και αντιμετωπίζω και εγώ στο έργο μου πολύ συχνά την ανάγκη αυτή να, λαμβάνω, να λάβω μια απόφαση εν γνώση του ότι ταυτόχρονα διατρέχουμε σημαντικό κίνδυνο οφείλω να πω ότι κατά την άποψή μου είναι πιο σημαντικό να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και να βοηθεί τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε δραματική κατάσταση αντί να κάθεται με άνεση και να αναμένει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες για να υπάρχει πλήρης ασφάλεια. Νομίζω ότι αυτό είναι και η άποψη του πολιτικού επίπεδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια ισορροπία που προσπαθούμε να αποκαθιστούμε διαρκώς ανάμεσα στο να είμαστε παρόντες στις καταστάσεις αυτές και ταυτόχρονα να σεβόμαστε την ανάγκη ελέγχου της δαπάνης των δημοσίων χρημάτων. Συχνά χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες εταίρων οι οποίοι βρίσκονται επιτόπου. Πολύ συχνά επίσης δεν είμαστε σε θέση εμείς να είμαστε ευθέως επί τόπου. Στις καταστάσεις αυτές οι κίνδυνοι είναι βεβαίως υψηλότεροι. Υπάρχουν χώρες όπου δεν μπορούμε καν να μεταβούμε εκεί και ο μόνος τρόπος για να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των αναγκών επισητιστικών, ε, ιατροφαρμακευτικών κλπ. των ντόπιων πληθυσμών είναι να δράσουμε μέσω διεθνών οργανισμών, μη κρατικών οργανώσεων, μέσω των υπηρεσιών τέτοιων ειδών εταίρων. Και αυτό κάνουμε. Και βεβαίως παρακολουθούμε διαρκώς που μεταβαίνουν τα χρήματα και αν τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τον σκοπό που, για τον οποίο μας, το έδωσε, μας τα έδωσε τα χρήματα αυτά ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος. Αλλά οφείλουμε να δεχθούμε τελικά ότι οι καταστάσεις αυτές ενέχουν περισσότερους κινδύνους από το να διεξάγει κανείς τις υποθέσεις του σε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον. Αυτή είναι όμως και η ουσία της δουλειάς μας. Μιλήσατε για την Παλαιστίνη, για την υπόθεση της Παλαιστίνης. Έχουμε εγκαταστήσει μηχανισμούς που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε πού μεταβαίνουν τα χρήματα. Και ωστόσο έχουμε καμιά φορά δυσκολίες, τα όσα έγιναν στην Γάζα για παράδειγμα, άλλαξε του όρους της βοήθειας και χρειάστηκε να προσαρμοστούμε. Και αυτό χρειάζεται χρόνο σε καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε βεβαίως. Αυτός όμως είναι ο κίνδυνος που εμπεριέχεται στην ίδια τη δράση και ελπίζω ότι η Επιτροπή σας θα αναγνωρίσει ότι οι δράσεις που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυσκολότερο να ελεγχθούν οι ορισμένε περιστάσεις. Και θα έλεγα πάλι καλά, και επιτρέψτε να το πω έτσι, που φτάνουμε σε ποσοστό σφάλματος 3%. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να μας καθησυχάσει, μας διασφαλίζει δηλαδή ότι είναι στο σωστό τρόπο με το οποίο χειριζόμαστε τα δημόσια χρήματα. Ο πρόεδρος Τόιρερ, ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε. Κοιτάξτε, δεν είναι και αλήθεια ότι από τη μια μεριά είναι οι ψυχροί βουλευτές και από την άλλη μεριά οι καλοί άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν. Για το θέμα της πολιτικής ανάπτυξης και της βοήθειας μπορεί να διαπιστώσει κανείς μετά από δεκαετίες αναπτυξιακής βοήθειας ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση πουθενά. Εγώ αυτό βλέπω στα 10 χρόνια που είμαι ευρωβουλευτή. Το ερώτημα τώρα σχετικά με την νομιμότητα. Όπως είναι φτιαγμένοι οι κανόνες και οι κανονισμοί και όπως δαπανώνται τα χρήματα μέσω επιδοτήσεων των προπολογισμών, δεν μπορούμε να μετρήσουμε αν τα χρήματα δαπανήθηκαν σωστά. Και ούτε εσείς άλλωστε μπορείτε να το πράξετε. Και αυτή ήταν και η έννοια της ανταλλαγής απόψεων με τον κύριο Πίνξτεν. Αυτό το τονίζω λοιπόν και πάλι, διότι αλλιώ προκαλείται η εντύπωση ότι εδώ είναι κάποιοι μικρόκαρδοι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν και την τελευταία δεκάρα. Όχι. Και μακάρι να ήμασταν ορισμένε φορέ, διότι θα ήταν και τα αποτελεσματά μα στην εξωτερική βοήθεια καλύτερα. Για το budget support, τι επιδοτήσει προπολογισμών, ο τρόπο που έγινε και παρά τι υποσχέσει από πολλών ετών και που θα γίνει και στο μέλλον, ο τρόπο αυτό οδηγεί στο ότι δεν γνωρίζουμε ποτέ τι πραγματικά επιτύχαμε. Θα αναμείνω με μεγάλο ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε του χρόνου πάλι γιατί δεν πέτυχε. Τουλάχιστον οι προκάτοχοί σας πάντοτε αυτό μας είπαν. Το μήνυμά τους ήταν πάντοτε αυτό. Δεν δέχομαι λοιπόν το υπονοούμενο ότι εδώ δήθεν κάθονται κάποιοι άνθρωποι άκαρδοι και άπονοι οι οποίοι κοιτάνε να ε, ελέγξουν και την τελευταία δεκάδα. Νομίζω, λέει ο Πρόεδρος, ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και όντως μπορώ να πω και εγώ ότι δεν έχουμε κακή ε, τύψη συνειδήσεως όταν ρωτούμε πού μεταβαίνουν τα χρήματα των φορολογουμένων. Στα κάτω της γραφής είναι και, αυτό, και αυτά μάλλον προϊόν κόπου και μόχθου. Και θέλουμε τα χρήματα που μας διαθέτουν οι φορολογούμενοι να φτάσουν πραγματικά στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Εμείς επικρίνουμε τη σπατάλη, την κατασπατάληση των χρημάτων, διότι τελικά αυτό επιβαρύνει τους ανθρώπους που χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Δεν βλέπω όμως να υπάρχει και καμιά αντίφαση μετά όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί κοινό πρέπει να είναι ο στόχος τα χρήματα να τα παρεχθούν σωστά και να καταλήξουν στους σωστούς δικαιούχους. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτού του θέματος της ημερησίας διατάξεως. Προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών έχει οριστεί η 26η Δευτέρου. Όπως είπα εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος αυτού και ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή καθώς και τους εκπροσώπους του Ελληνικού Συνεδρίου. Okay, dann kommen wir zu den äh, anderen Institutionen, other institutions. Wir haben hier zwei. Äh, κύριε, ε, έχουμε τώρα δύο ε, εισηγητές, Τάμας Ντόιτς και Μπογκοσλαβ Σόνικ, που δεν τον έχω δει ακόμη. Α, η κυρία Γκρέσλι τον εκπροσωπεί, τον Σόνικ. Σε ποιον να δώσω πρώτα το λόγο, στο ελεγκτικό συνέδριο ή θέλετε εσείς πρώτος κύριε Ντόιτς. Εσείς, κύριε Ταμάς, Deutsch. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Έχω αναλάβει την έκθεση για την, εξωτερική υπηρεσία, για την υπηρεσία εξωτερικής δράσεως στο Ελεκτικό συνέδριο και το δικαστήριο για, τον... για την εκτέλεση των προπολογισμών τους δεν βλέπω ουσιαστικά ουσιώδη σφάλματα Μόνο ως προς τις ε, διοικητικές δαπάνες έχει κάνει το ελεκτικό συνέδριο κάποιες παρατηρήσεις για την υπηρεσία εξωτερικής δράσεως. Και θα ήθελα για τις εκθέσεις αυτός, αυτές να πω ότι η Επιτροπή μας έχει Κατα... έχει υποβάλει 47, 54 και 234 ε, ερωτήσεις προς τα τρία αυτά όργανα, έλαβε 338 απαντήσεις στις αρχές του χρόνου μας έστειλαν τις απαντήσεις τους τα όργανα αυτά, συμβάλλοντας έτσι στην ε, αποτελεσματική υλοποίηση του έργου μας και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους και των τριών ε, οργάνων που τήρησαν πάνω απ' όλα τα πολύ αυστηρά χρονικά περιθώρια. Λάβαμε πριν από δύο εβδομάδες τους εξολογισμούς της ετήσιας χρήσης και εδώ βλέπουμε τις πιο σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων με τα κύρια ποσά, με τα επιμέρους ποσά. Θα περάσω τώρα στα επιμέρους όργανα και ξεκινώ με το δικαστήριο. Ευρωπαϊκό δικαστήριο λοιπόν. Το 2012 το το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε, δεσμε, έχει πιστώσει υποχρεώσεων 343 εκατομμύρια. Η εκτέλεση ήταν στο 98,5%. Σχετικό επίσης βλέπουμε ότι το δικαστήριο του 2012 ολοκλήρωσε, πραγματοποίησε την ιστορική του μεταρρύθμιση με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο δικαστήριο. Διότι το κύριο ζήτημα εδώ είναι το πρόβλημα των εκρεμών δικών. Είναι ακόμη πολύ ψηλό ο αριθμό των εκρεμών δικών ενώπιον του δικαστηρίου και άρα αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που καλείται να επιλύσει το το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και ναι μεν κατατίθενται περισσότερες προσφυγές χρόνο με το χρόνο, αλλά και οι διαδικασίες είναι μακροχρόνιες. Περιμένουμε λοιπόν να μειωθεί με επιτάχυνση των διαδικασιών μετά τη μεταρρύθμιση το 2013 σχέση με το 2012 ο αριθμός των εκκρεμών δικών. Πάντως η τάση μέχρι το 2012 ήταν ανωδική σε σχέση με το 2011. Από 849 σε 886 εκκρεμείς δίκες και λιγότερο ε, λιγότερος αριθμός των δικών που είχαν ε, ολοκληρωθεί. Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι μεγάλο μέρος του προσωπικού, το μισό σχεδόν προσωπικό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, απασχολείται στη μετάφραση, είναι μεταφραστές. Η πολυγλωσία έχει και ε, στην πράξη εξασφαλιστεί και στην ε, ακροαματική διαδικασία. Και αυτό βέβαια εξηγεί και το μεγάλο αριθμό μεταφραστών αλλά και διερμηνέων που εργάζονται για το δικαστήριο. Πράγμα το οποίο συνεπάγεται και σημαντική διοικητική ε, επιβάρυνση αλλά και σε κόστος, μεγαλύτερες δαπάνες. Το δικαστήριο προσπαθεί να μειώσει όμως και σε αυτό το σημείο το κόστος. Το επόμενο μας όργανο είναι το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο επαληθεύει την εκτέλεση των λογαριασμών των ευρωπαϊκών οργάνων. Εξωτερικός ελεγκτής είναι αυτός ο οποίος επαληθεύει τον ισολογισμό του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και μας λέει ότι για το 2012 καταγράφεται θετική εικόνα για το ελεγκτικό συνέδριο. Οι πιστώσεις υποχρεώσεων ήταν 137 εκατομμύρια ευρώ για το 2012 με ποσοστό απορρόφησης μεγαλύτερο από 96%. Για τις ειδικές εκθέσεις. Το χρονικό περιθώριο που απαιτείται για την εκπόνησή τους περιορίστηκε στους 20 μήνες. Ο στόχος όμως των 18 μηνών που είχε οριστεί δεν έχει επιτευχθεί ακόμη για την εκπόνηση, ολοκλήρωση και κατάθεση ειδικών εκθέσεων. Το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει για το ελεγκτικό συνέδριο να σημειώσουμε για τη λειτουργία του και το κόστος λειτουργίας ότι είναι πολύ μεγάλες οι αποκλήσεις στο κόστος μετάφρασης ανασελίδα ανάλογα με τις γλώσσες. Αυτό έχει να κάνει και με μεθοδολογικούς παράγοντες. Γιατί μερικές φορές μπορεί να καταγραφεί το κόστος μετάφρασης μία δαπάνη ενώ κάποιες άλλες όχι. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα μεθοδολογίας και ανάλογα με τη μεθοδολογία αυτή διαφοροποιείται η τιμή ανασελίδα για την μετάφραση. Στο δικαστήριο παραδείγματι. Στο κλείσιμο των λογαριασμών έχουμε κατά σελίδα 98 ευρώ κόστος. Ενώ για το δικαστήριο, για το ελεκτικό συνέδριο 246 ευρώ η σελίδα Αυτό, όπως είπα, έχει να κάνει με τη μεθοδολογία που επιλέγεται για τον υπολογισμό αυτού του κόστους. Ε, πάντως, πιστεύω το επόμενο έτος θα πρέπει να έχουν ε, τα, τα, τα, όργανα όλα έναν ομοιόμορφο τρόπο υπολογισμού του κόστους ε, για τη μετάφραση της ε, σελίδας, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες οι, συγκρίσιμα τα μεγέθη και να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν ανομαλίες ως προς την, ως προς την δαπάνη. Επίσης πρέπει να βελτιωθεί η συμμόρφωση στις εργασίες του συνεδρίου ε, έναντι των πολιτικών προτεραιοτήτων που ορίζει το Κοινοβούλιο. Ανάλογα λοιπόν με τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου θα πρέπει το ελεκτικό συνέδριο να προσαρμόσει το πρόγραμμα εργασίας του. Το 2012 παρέπεψε 16 υποθέσεις στην Όλαφ, το ελεγκτικό συνέδριο, με υποψία απάτης. 12 ανακριτικές διαδικασίες ξεκίνησαν, για τις οποίες δεν έχουμε λάβει ενημέρωση. Δεν ξέρουμε δηλαδή πόσες περιπτώσεις έχουν παραπευθεί από ευρωπαϊκά όργανα, σε πόσες έχουν ξεκινήσει ανακριτικές διαδικασίες και τι είδους ε, αποτέλεσμα προκύπτει από τις έρευνες της Όλαφ, εάν ξεκίνησαν. Εδώ, ακόμη και με την ε, δεδομένη προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε σε ποιε περιπτώσεις η Όλαφ κάνει έρευνες και τι είδους αποτέλεσμα προκύπτει από αυτές. Και ολοκληρώνω με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ένα όργανο ε, με μεγάλη έκταση, 7.000 υπαλληλούς Δεν θέλω να αναφερθώ λεπτομερώς στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο αριθμό των ε, εργαζομένων στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Πάντως εν γέννη βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα προπολογισμό άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ και ποσοστό εκτέλεσης άνω του 99%. το ελεκτικό συνέδριο έχει κάνει μόνο μία παρατήρηση σε σχέση με την υπηρεσία εξωτερικής δράσεως για τον τρόπο λειτουργία γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με τις ε, δαπάνε για κοινωνικέ παροχέ που έχουν ε, ε, εγγραφεί στον προπολογισμό. Ένα ερώτημα το οποίο είχε διατυπωθεί ήδη από την προηγούμενη χρονιά και είχαμε ζητήσει να υπάρξει ένα σύστημα κοινωνικές παροχές όπως οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα τέκνων κτλ. να μην καταβάλλονται εις διπλούν στον εργαζόμενο, δηλαδή και από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και από τους Εθνικούς Προϋπολογισμούς. Είναι θέματα τα οποία ασφαλώς ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα. Για τις γραπτές μας ερωτήσεις. η συζήτηση που ολοκληρώθηκε με αυτή την γραπτή ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων δείχνει ότι η υπηρεξία εξωτερικής δράσεως έχει ψηλές ε, δαπάνες. Σφάλματα σημαντικά δεν έχουμε δει. Το 2012 ωστόσο βλέπουμε ότι η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία ε, υστερεί αρκετά. Περισσότερο δεν θέλω να επεκταθώ στο θέμα αυτό. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω ότι εν όλο 514 υπάλληλοι της ε, υπηρεσίας αυτής βρίσκονται στην βαθμολογία Α12 ή άνω. Έχουν μισθούς υψηλούς με συνολικό ποσό για τους 514 αυτούς υπαλλήλους, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Πέραν αυτών, αυτοί οι υπάλληλοι ε, έχουν και άλλες παροχές πέραν των μισθών τους. Και επίσης 3.360 υπάλληλοι, λεγόμενοι local agents, οι επιτόπου ε, απασχολούμενοι της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης έχουν συνολικά συνολικές αμοιβέ ανώτερες των 3.000 ευρώ. Ο καθένας χωρίς λοιπόν να θέλω να γίνω σαρκαστικός την σήμερον ημέρα και στον κόσμο που ζούμε Είτε πρόκειται για την Ουγγάντα είτε πρόκειται για τη Βολιβία. Υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, υπάλληλοι οι οποίοι κατά μέσο όρο εισπράττουν 3.074 ευρώ το μήνα ως μισθό. Πράγμα το οποίο για τις χώρες αυτές μου φαίνεται δυσανάλογα υψηλή αμοιβή. Ο αρμόδιος γενικός διευθυντής, όταν τον ρωτήσαμε, μας είπε ότι υπάρχουν ακόμη και υψηλότερες αμοιβέ σε ορισμένες περιοχές του κόσμου. Δηλαδή είναι μάλλον μέσο όρο αυτό που βλέπουμε. Μια μεσαία κατηγορία αυτό που αναφέρω. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει δυνατότητα ασφαλώς να οργανωθεί η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας με πιο οικονομικό τρόπο. Ένα άλλο θέμα πάλι από παρατήρηση και για το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, είναι η, η γεωγραφική κατανομή. Τα 13 κράτη τα οποία εντάχθηκαν τα τελευταία δεκαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν ε, υποεκπροσώπηση. Έχουμε 131 ε, αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο και μόνο 30 εξ αυτών έχουν επανδρωθεί από διπλωμάτες των 13 νέων κρατών μελών για την ε, κτηριακή υποδομή και τη σχετική πολιτική της ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης πάλι υπάρχουν ερωτήματα, ερωτηματικά. Δεν λάβαμε σε όλες μας τις ε, γραπτές ερωτήσεις επαρκής και ικανοποιητικέ απαντήσεις. Και συνεχίζουμε τις επαφές. προκειμένου να διευκρινίσουμε τα ακόμη εκρεμή ζητήματα. Για να συνοψίσω κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πέραν των ε, ποσών και των προβλημάτων που επεσήμανα, προτείνω να χορηγηθεί η απαλλαγή, διότι τα μεγέθη για τα οποία μιλούμε δεν έχουν να κάνουν με αποτελεσματικότητα, μάλλον τα μεγέθη για τα οποία μιλούμε έχουν να κάνουν περισσότερο με αποτελεσματικότητα στη λειτουργία, αλλά όχι με την νομιμότητα ή, το, την τήρηση των κανόνων για την εκτέλεση των λογαριασμών αυτών των οργάνων. Έχουν εκτελέσει τους προϋπολογισμούς τους τα όργανα αυτά κατά τρόπο σωστό, ε, νομότυπο και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να μην τους χορηγηθεί η απαλλαγή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και το δικαστήριο και το Ελεκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση, τη Γραμματεία της Επιτροπής του Ελέγχου του Προπολογισμού, ε, όλους βέβαια τους συναδέλφους που με, βοήθησαν και με υποστήριξαν επικοδομητικά σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 25 Φεβρουαρίου. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία στις 18 Μαρτίου να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας για να περάσει η έκθεση στην, στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Και περιμένω τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Άκουσα ότι τώρα εσείς εκπροσωπείτε τον κύριο Σόνικ. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ο κύριος Σόνικ κολλείεται σήμερα, αλλά θα σας αναπτύξω ε, τα σχόλιά του εγώ. Και πρώτα ο κύριος Σόνικ ευχαριστεί τα θεσμικά όργανα για τη συνεργασία τους και για την διαβίβαση των σχετικών πληροφοριακών ε, στοιχείων και τη συναντήσεις με τους ευρωβουλευτές. Δεν σημειώνονται μείζωνα προβλήματα. Φέτος δεν σημειώθηκαν ουσιαστικά σφάλματα και τα, τα ποσοστά σφαλμάτων βελτιώθηκαν από πέρσι. Ο κ. Σόνικ εκφράζει την ικανοποίησή του για την καλή λειτουργία της συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής Περιφερειών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και σημειώνει και τον οικονομικό χαρακτήρα τον ορθό οικονομικό χαρακτήρα της εργασίας της ε, Επιτροπής των Περιφερειών και με την απαραίτητη ενημέρωση, ιδίως ό,τι αφορά τη, τα, τα, τις προφορίες σχετικά με τα επιδόματα ταξιδιού, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα παλαιότερα. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο. Δυστυχώς ο κ. Σόνικ εδώ δεν μπορεί να πει το ίδιο. Η συνεργασία με το Συμβούλιο δεν είναι τόσο ομαλή όσο θα ήθελε να δει ο ίδιος ο κ. Σόνικ, το Συμβούλιο εξακολουθεί να αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου και δεν προσέρχεται και ώρας να προσκαλείται. Η στάση του αυτή αποδεικνύει ότι το Συμβούλιο δεν σέβεται την λειτουργία ελέγχου του προεπολισμού του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό ο εισηγητής διαβίβασε τις ερωτήσεις που απίθυνε κανονικά στο Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία απήντησε με επιστολή από 23 ε, Ιανουαρίου. Ο κ. Σόνικ σημειώνει ότι η απάντηση της Επιτροπής λέει ότι δεν απαντά για λογαριασμό του Συμβουλίου για να μην αναμειχθεί σε εσωτερικά θέματα του θεσμικού αυτού οργάνου. Σημειώνει όμως ότι όλα τα θεσμικά όργανα είναι υποχρεωμένα να συνεργάζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα απαλλαγής. Με την συμβολή της ελληνικής αντιπροσωπείας, το ε, μόνιμης αντιπροσωπείας δηλαδή, το Συμβούλιο θα ιδρύσει ε, ομάδα εργασίας η οποία θα εγκύψει το θέμα. Βέβαια, όταν δεν χορηγούνται σχετικές πληροφορίες, δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να θεμελιώσει απόφαση για τη χορήγηση της απαλλαγής. Και γι' αυτό ο εισηγητής προτείνει αναβολή της χορηγήσεως της αναβολής στο Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, λέει, θα πρέπει να καταδείξουμε την κατεύθυνση προς το μέλλον και γι' αυτό ο εισηγητής προτείνει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας καθώς και ακρόαση ή εργαστήριο που να ε, συζητήσει μια νομική ανάλυση της καταστάσεως και με ενδεχόμενη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή να ζητήσει διασάφηση των ε, διατάξεων της συνθήκης. Ο κύριος Σόνικ αναμένει τα σχόλιά σας και σημειώνει ότι η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι η 25η Φεβρουαρίου και αυτά κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σάβαμη. Υπάρχουν ερωτήσεις. Εσείς κύριε Γκάιερ. Ναι κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Που είναι και η πιο σημαντική βέβαια. Εγώ συμφωνώ με την στάση του εισηγητού που προτείνει αναβολή της απαλλαγής Θα συστήσω όμως μια διαφορετική προσέγγιση. Νομίζω ότι έχουμε νομικά την δυνατότητα σε ό,τι αφορά πρωτοβουλίες που ενδέχεται να αναλάβει η παρούσα Επιτροπή τις οποίες μέχρι τώρα δεν έχουμε δοκιμάσει επαρκώς. Και νομίζω η σχετική εργασία πρέπει να γίνει στις πολιτικές ομάδες που να εμπαθύνουν στο ερώτημα ανεξαρτήτως αναβολής απαλλαγής στο ερώτημα αν υπάρχει πολιτική πλειοψηφία για την καταγγελία της περίφημης Συμφωνίας Κυρίων τουλάχιστον στα έγγραφα που έλαβα εγώ από το Κοινοβούλιο όταν έγινα εδώ Ευρωβουλευτής προπενταετίας τα χαρτιά αυτά έλεγαν, αν και ο κύριος Όντριγκας λέει ότι δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, για μια συμφωνία κυρίων. Και ο πυρήνα τη συμφωνία κυρίων ήταν ότι δεν αγγίζουμε ημέν του προπολογισμού των δε μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αν θέλουμε να το πράξουμε αυτό, ω ελεγκτικό συνέδριο δηλαδή, αυτό βέβαια μόνο οι πολιτικέ ομάδε μπορούν να το αποφασίσουν γιατί τότε βέβαια πρόκειται για ανοιχτή πολιτική σύγκρουση. Και επιτιθέμεθα τότε κατά του Συμβουλίου και λέμε ότι ως Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού ερχόμαστε και ελέγχουμε τον προϋπολογισμό σου. Τότε θα κάνουν και οι ίδιοι το ίδιο για μας. Άρα είναι δίκοπο μαχαίρι και χρειάζεται προσοχή. Δεύτερη επιλογή που λίγο πολύ το ανακοίνωσε ο Πέτρι ως εκπρόσωπος του εισηγητή, είναι προσφυγή στο δικαστήριο. Εμείς έχουμε σχετικό λόγο, αυτό θεωρώ. Και η τελευταία ακρόαση, αυτό κατέδειξε διότι και οι τρεις εμπειρογνώμονες που είχαμε προσκαλέσει συμφώνησαν ότι τουλάχιστον η πρόσβαση στα έγγραφα είναι κάτι που πρέπει να χορηγηθεί στο Κοινοβούλιο. Αν όμως προσφύγει το, δικα... το κοινοβούλιο στο δικαστήριο, τότε θα πρέπει να είναι απόφαση του συνόλου του Κοινοβουλίου και όχι μόνο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Εγώ είμαι διατεθειμένο να προχωρήσω προ την κατεύθυνση αυτή και να κάνω και τη σχετική εργασία στην πολιτική μου ομάδα. Όμω τότε θα πρέπει να το κάνουμε όλοι. Τουλάχιστον όλε και όλοι όσοι θέλουμε να διατηρήσει το όργανο τα δικαιώματά του. Και θα πρέπει τότε να εξετάσουμε με τον κατάλληλο τρόπο εάν υπάρχει ενδεχόμενο να μας υποστηρίξουν οι πολιτικές μας ομάδες. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε νομίζω εύκολο είναι να ζητήσουμε από την νομική μας υπηρεσία να μας προτείνει την κατάλληλη διαδικασία για να καταλήξουμε σε μια, όπως ελπίζω, θετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όμως αυτό νομίζω ότι δεν απαιτεί καμία παραπέρα διαδικασία μέσα στα πλαίσια της ίδια της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, θα πρέπει απλά να στραφούμε στις πολιτικές μας ομάδες και να τους ζητήσουμε την υποστήριξη τους. Ευχαριστώ. Είναι και Γκρέσλε. Κοιτάξτε, συμφωνία κυρίων, εάν υπάρχει τέτοια τότε μάλλον πρόκειται για μονομερή δήλωση του Συμβουλίου. Απομένως εδώ χρειάζεται κάποιος διαχωρισμός. τα όσα προτείνει ο Σόνικ είναι να σκεφτούμε ότι αν καταλήξουμε σε αναθεώρηση της συνθήκης, γιατί κάθε στιγμή θα καταλήξουμε εκεί, θα πρέπει να είναι σαφές ότι και το θέμα αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Άρα θα χρειαστούμε μια ξεκάθαρη διατύπωση. Και αυτή η διατύπωση πρέπει να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας, που πάει να πει ότι πρέπει να συμμετάσχει η Επιτροπή Συνταγματικών και ούτω καθεξής. Άρα το νέο Κοινοβούλιο θα πρέπει να σκεφτεί εάν ίσως μαζί με την ΑΦΚΟ να κάνει μια προσπάθεια να εκπονήσει ένα νέο άρθρο γιατί πρόκειται για ένα κάρφος εν του οφθαλμό μας το οποίο έχουμε εδώ και χρόνια και μας πονά και μας ενοχλεί και ίσως είναι δυνατό να το επιτύχουμε. Χρειάζεται λοιπόν προετοιμασία εγώ τηλεφώνησα στον Έλληνα πρέσβη, ο οποίος καταβάλει προσπάθεια και πάλι να ρυθμίσει το θέμα. Αλλά όσο από το Συμβούλιο δεν λαμβάνουμε απολύτως κανένα σημάδι, Βεβαίω να μιλεί κανεί είναι δυνατόν. Εδώ και δέκα χρόνια εγώ μιλώ και μιλώ και ξαναμιλώ με το Συμβούλιο. Ουδεμία πρόοδο. Διότι το κρίσιμο θέμα, δηλαδή αν επιτρέπεται οι κυβερνήσεις να ελέγχουν ένα κοινοβούλιο, εγώ πιστεύω πως όχι, σαφώς. Όμως οι κυβερνήσεις έχουν άλλη άποψη βέβαια. Βεβαίω, στι χώρες τους ποτέ δεν θα τολμούσαν να αγγίξουν τη Βουλή τους. Εδώ στις Βρυξέλλε βεβαίως θεωρούν ότι μπορούν. Από άποψη του Κοινοβουλίου δεν είναι δυνατόν όμω να μα ελέγχουν οι κυβερνήσει. Πάντω, όσο δεν σημειώνεται καμιά πρόοδος δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να προχωρήσουμε σε νέες πρωτοβουλίες. Εγώ έχω κουραστεί πια να θέτω το θέμα σε κάθε νέα Προεδρία του Συμβουλίου. Και οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων ας σκεφτούν τι εικόνα θα δώσουν προς τα έξω. Να θέλουν να βγουν και να πούν στον ψηφοφόρο ότι έχει σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά οι κυβερνήσεις θέλουν να το ελέγχουν. Τι εικόνα είναι αυτή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο Μούλτερ. Η κατάσταση με το Συμβούλιο κάθε χρόνο επαναλαμβάνει τα ίδια επιχειρήματα. Πριν φτάσουμε στο δικαστήριο, ίσως μπορούμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, να κηρύξουμε τη λήξη της Συμφωνίας Κυρίων. Αυτό νομίζω, καθώς η θέση του Κοινοβουλίου είναι ισχυρότερη σε σχέση με την απαλλαγή, διότι η τελική απόφαση, όπως ορίζει η συνθήκη, είναι στα χέρια του Κοινοβουλίου. Άρα, τι μας ε, υποχρεώνει να διατηρήσουμε ενίσχυα τη Συμφωνία Κυρίων. Εγώ σκέφτομαι να καταθέσω και σχετική τροπολογία. Και βλέπουμε. Τη δέχεται το Κοινοβούλιο ή δεν τη δέχεται. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ίσως ήταν ευφυές από πλευράς της Προεδρίας της ώστε ότι καθόμαστε σε, ότι επιλέγει αυτή η αίθουσα γιατί καθόμαστε γύρω-γύρω από ένα κύκλο όλοι μας και ίσως είναι καλό τώρα να αναλογιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο εισηγητής μέσω του εκπροσώπου του μας προτείνει μια έκθεση πρωτοβουλίας, μια λύση πρακτική και ρεαλιστική έκθεση η οποία θα επιτρέψει την διαμόρφωση της θέσεως του Κοινοβουλίου, αλλά βέβαια θα πρέπει και οι συνάδελφοι να αναλογιστούν τι θέλουμε να ζητήσουμε εμείς ως Κοινοβούλιο. Και εν προκειμένου το το ερώτημα, εάν αποκλίνουμε από τη μέχρι τώρα θέση μας ή αν αξιοποιούμε τη δυνατότητα τουλάχιστον για την υποβολή ερωτήματος στο δικαστήριο. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να ζητήσουμε από το, να προτείνουμε στο Κοινοβούλιο να απευθυνθεί στο δικαστήριο με μια έκθεση πρωτοβουλία, να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο και ίσω ε, εναλλακτικά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και τη δυνατότητα να προσκληθούν και 28 Υπουργοί των Οικονομικών ε, σε μια συνεδρίαση ή να σκεφτούμε και άλλες λύσεις κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, γιατί η εντύπωση που έχω μέχρι τώρα είναι ότι άλλα τμήματα του Κοινοβουλίου δεν δείχνουν το ίδιο ε, ενδιαφέρον, δεν αποδίδουν τόσο μεγάλη σημασία δηλαδή στην απαλλαγή του Συμβουλίου. Για μας όμως είναι πολύ σημαντικό. Είναι ζήτημα δημοκρατικού ελέγχου και ίσως καλό θα είναι να αναλογιστούμε αν μπορούμε σε μια έκθεση πρωτοβουλίας να συμπεριλάβουμε τοποθετήσει, διεκδικήσει που δεν είναι απλώς μια έκκληση προς το Συμβούλιο, αλλά κάτι πιο ουσιαστικό. Κύριο κύριος Γκάιερ. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ που το διευκρινίζεις και το παραλαμβάνεις, Ίγκε. Ασφαλώς έχει νόημα το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και να τοποθετηθεί. Για την έκθεση πρωτοβουλίας πάντως θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί Γιατί και με αυτά που είπε τώρα, Μιχαήλ, μην ξεχνάμε τις παράπλευρες απώλειες, τις πολιτικές παράπλευρες απώλειες που μπορεί να είναι πολλαπλές και πολλοί επίπεδες. Ας αναλογιστούμε λοιπόν τι θέλουμε όλοι μας, τι θέλουν διάφορες πολιτικές ομάδες, τι είδους διαφορετικές επιλογές έχουμε, τι είδους πολιτικές ε, έχουμε και πλειοψηφίε. Ίσως τελικά δηλαδή να μην φτάνουν αυτές οι ισορροπίε και πλειοψηφίε για να διατυπωθεί μια σαφή ε, θέση του Κοινοβουλίου και ω εκ τούτου θα προτιμούσα να μην υπάρξει ε, έκθεση πρωτοβουλία. Άρα θα πήγαινα προ μια αναλλακτική ή προ μια έκθεση πρωτοβουλίας η οποία απλώς ε, αναφέρει διαφορετικές επιλογές. Δεν μας βοηθάει αυτό πάντως σε μια γενικότερη πολιτική συζήτηση, γιατί ενδέχεται να χαθεί η ουσία της συζήτησης μέσα στο διάλογο των πολιτικών ομάδων, να φτάσουμε στην Ολομέλεια και να προχωρήσει η συζήτηση μέσα από πολιτικό, πολιτικές πιέσεις, στρατηγικές πιέσεις και στη δε Ολομέλεια να έχουμε αποτελέσματα που δεν τα περιμέναμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να εξυπηρετεί τον κοινό στόχο, αλλά με όσο δυνατόν λιγότερε παράπλευρε απώλειε. Το Συμβούλιο είναι παρόν. Μπορούμε νομίζω να αναλογιστούμε τι είδου λύσει έχουμε για την κλιμάκωση τη πίεση. Ε, νομίζω ότι η ιδέα αυτή να προσκαλέσουμε 28 υπουργού των οικονομικών ε, θα καταλήξει μάλλον σε 28 αρνητικές απαντήσεις από τους υπουργούς των οικονομικών, άρα ίσως να μην ε, είναι πολύ πρόσφοροι. Η άλλη λύση, το επόμενο βήμα θα ήταν να γίνουν οι συνεδριάσεις και να δείξουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε στην ουσία στο κύριο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Εάν θεωρούν πάντως οι πολιτικές ομάδες ότι είναι σημαντικό να τοποθετηθούν στο θέμα αυτό και οι επικεφαλής των εκλογικών τους ληστών και να ασκήσουν την πολιτική πίεση, τότε ίσως μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστικό θέμα πολιτικού διαλόγου το ζήτημα αυτό και να προχωρήσει. Βέβαια είναι σημαντικό να προχωρήσει η συζήτηση στο Κοινοβούλιο με ουσία. Να μην αφήσουμε δηλαδή να χαθεί στον υπολογισμό της ημερήσιας διάταξης. Είναι κάτι το σημαντικό. Μπορούμε να δούμε αν υπάρχει υποστήριξη από τα κράτη-μέλη και από τα εθνικά κοινοβούλια ίσως όπου θα ήθελα να πω ξεκάθαρα πως ε, για τον έλεγχο που ασκεί το Κοινοβούλιο στα ε, μέλη του Συμβουλίου, δηλαδή εθνικές κυβερνήσεις, υπάρχουν σημαντικές επιφυλάξεις. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε εάν η εναλλακτική, η επιδίωξη μιας τροποποίησης της συνθήκης κατά τρόπον ώστε να μπορούν να ελέγχουν το Συμβούλιο τα εθνικά κοινοβούλια, που είναι ίσως μια λύση πιο ευχάριστο συμβούλιο, γιατί έτσι ως συνομοθέτη στο Συμβούλιο δεν θα εκτίθεται στον έλεγχο του, του άλλου, του έτερου συνομοθέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή, αλλά από τα εθνικά κοινοβούλια, είναι κάτι το οποίο ίσως οι εθνικοί βουλευτές ενδιαφέρονται να το δουν. Το θέμα είναι αν εμείς θεωρούμε ότι έχουμε αρκετές δυνάμεις ώστε να εντείνουμε τις πιέσεις και αν μπορούμε να σταθούμε στο ύψος αυτών των ε, περιστάσεων σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα και κυρίως με το Συμβούλιο και αν μπορέσουμε να φέρουμε τους αρχηγούς κρατών και συζητήσεων να συζητήσουν τα θέματα αυτά, ίσως και με, την, ε, με το προσωπικό τους κύρος και την πολιτική τους εμβέλεια οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων να μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτής της θεματολογίας ε, στα κράτη-μέλη. Αυτές είναι κάποιες ιδέες. Είμαι πάντα στη θέση σας βεβαίως, εάν αποφασίσουμε να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Πάντως, θεωρώ ότι ναι είναι καλό να τοποθετούμαστε ξεκάθαρα και να λέμε τι εννοούμε και τι θέλουμε, αλλά από την άλλη πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και αν προωθούμε μία λύση, να ξέρουμε ότι αυτή η λύση θα έχει τη στήριξη της πλειονοψηφίας του Κοινοβουλίου. και ότι μπορεί να υιοθετηθεί και να προωθηθεί από τον μελλοντικό πρόεδρο ή την μέλουσα πρόεδρο του Κοινοβουλίου έναντι του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Θέλω απλά να σας ενημερώσω ότι θα διαβιβάσω στον κύριο Σόνικ τις σημειώσεις που ε, έχω καταγράψει από αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να στέκανε άλλο το λόγο. Ούτε από την Επιτροπή βλέπω να στέκανε το λόγο. Αυτή τη στιγμή. Άρα κλείνουμε και το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης και εάν διαβάζω σωστά και την ημερήσια μας διάταξη. Γιατί συνεχίζουμε με τους συντονιστές. Τελειώνει λοιπόν εδώ το δημόσιο μέρος της συνεδριάσεως. Αύριο θα συνεχίσουμε, αύριο το πρωί. Και περνάμε στις συνεδρίες και κλεισμένων των θυρών.